Ladies and Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Ξεκινήσει η συνεδρίαση, είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι. Που καλωσορίζω τον στρατηγό Ζαν Πολ Παλομερός. Ανώτατο διοικητή ΝΑΤΟ από τον Ορφόλκ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τις ιδέες του για την ε, μεταμόρφωση της μαχικής διοίκησης ύστερα από την σχετική συνεδρίαση μια σημαντική ευκαιρία με πολλές και σημαντικές αποφάσεις επιτρέψτε μου λοιπόν να σας ενημερώσω για τις σημερινές διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την ενημέρωση. για την ε, μεταμόρφωση της ε, συμμαχικής διοίκησης της που Ουαλίας, ο κύριος Παλομερός και στη συνέχεια η κυρία Κλωτ Φρανς Αρνού επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας. Κάπου στις 4 θα μας έρθει για να μας δώσει και εκείνη την πλευρά της προτάσεις και ιδέες για το ευρωπαϊκό δυναμικό μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και εν ώψη της επερχόμενης Συνοδού των Βρυξελών τον Ιούνιο του 2015. Στόχο έχει να επεξεργαστεί θέματα της ΚΕΠΑ. Θέλω λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο και για άλλη μια φορά να καλωσορίσω τον στρατηγό Παλομερός ε, και να του δώσω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Μιλώντας γαλλικά θα ξεκινήσω. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας εδώ. Χαίρομαι που είμαι για δεύτερη φορά μαζί σας γιατί ήδη πριν από ένα χρόνο είχα έρθει και θα ήθελα να λάβω το λόγο ακριβώς ε, σε αυτές τις ιδιαίτερα πυκνές ανταλλαγές που συμβαίνουν από τους εκπροσώπους ε, με, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ η κυρία Μαγκερίνη είναι η Γενική Γραμματέας ε, και έδωσε μια κοινή συνέντευξη τύπου που έκανε ιδιαίτερη καλή εντύπωση τώρα τελευταία και η κυρία Μογκερίνη επίσης ε, χθες ε, ήταν παρούσα στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ έλαβε το λόγο και νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Επίσης αυτή τη στιγμή Έχουμε μια περίοδο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2013 και στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ θα μιλήσω για την Ουαλία σε λίγο. Βλέπουμε την αναλλαγή αυτή και όπως το επενθυμίσατε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά το 2015. Άρα λοιπόν ε, υπάρχει μια αρέουσα δυναμική και θέλουμε αυτή να έχει την καλύτερη δυνατή συνοχή. Οι δύο οργανώσεις ε, βασίζονται σε 22 κράτη που συμμετέχουν ε, και μπορούν να γνωρίσει ακριβώς ότι υπάρχει μια ε, συμπληρωματικότητα όσον αφορά τη δράση του σε περιπτώσεις κρίσης και θα ήθελαν να, αυτή την εργασία να τη συνεχίσουν με πολλαπλές προσπάθειες για να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και τα κράτη αυτά και στη, για θέματα δαπανών άμυνας κοινής ενέργειας λοιπόν και από πολιτικής πλευράς υπάρχει μια όθηση εσείς την εκπροσωπείτε αυτή την πολιτική όθηση επίσης μια στενή στρατιωτική συνεργασία στα πολιτικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί ένα μεγαλύτερο άνοιγμα όπως και διαφάνεια μεταξύ των δύο αυτών οργανώσεων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ρεαλιστές πρέπει να είμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν ε, σημαντικές κοινέ προκλήσεις. Απαιτούνται απαντήσεις ε, συλλογικές και συμπληρωματικές ε, για την ειρήνη, την ασφάλεια στην Ευρώπη χρειάζεται μια ατλαντική κοινή προσπάθεια και ένας καλύτερη ισορροπία όσον αφορά τις δαπάνες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα. Και οι προοπτικές αυτές έχουν να κάνουν με τις προσπάθειες αυτές μεταρρύθμισης εδώ και στο νότο στρατηγείο που βασίζεται στις ΗΠΑ, στο Norfolk ε, είναι ο πυλώνας ακριβώς ε, που βασίζεται ε, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό σύντομα. Από το ξεκίνημα πριν από 10 χρόνια, το 2003, προσπαθούμε να ε, ρυθμίσουμε την προσαρμογή του ΝΑΤΟ και για τις περισσότερες δυνατότητες στρατιωτικές, ε, εξοπλισμός που έχει να κάνει με αυτό, αλλά και την όλη απασχόληση, την οργάνωση, την ε, οργάνωση ακριβώς, τις ασκήσεις κλπ. Αλλά λοιπόν προσαρμογή και ασκήσεις για το μέλλον και αυτό με την καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή προπαρασκευή να μπορέσουν να υπάρξει μια κατάλληλη συνεργασία ανάμεσα στις ε, συμμαχικές δυνάμεις και με τους εταίρους μας όλα και περισσότερο. Και όλα αυτά βασίζονται σε ένα συλλογισμό για πώς θα είναι το μέλλον που αυτό μας απασχολεί σχετικά με αυτή τη μεταρρύθμιση να προετοιμάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σχεδιάσουμε το μέλλον. Η μεταβολή αυτή είναι διαρκής διαδικασία και με συμβατικές αλλά και με πυρηνικές δυνάμεις να είναι αξιόπιστες για να ανταποκριθούν ακριβώς στην αντίληψη του ΝΑΤΟ όπως υπόθηκε στην Σαβόνα, τη διαχείριση κρίσεων, τις δαπάνες και τη συνεργασία. Όπως το είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, εδώ οι δύο οργανώσεις αντιμετωπίζουν δύο κοινέ προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα, αντιμετωπίζουμε κάτι το περίπλοκο και που μεταβάλλεται συνεχώς ε, όσον αφορά τα ε, σύνορα της Ευρώπης. Στην Ουκρανία η κρίση εκεί βλέπουμε μια ευρυδική νέα κατάσταση και χρειάζεται να ε, στρατιωτικές, προστρατιωτικές, ε, πολιτικές, συμβατικές λοιπά δυνάμεις να μπορέσουν να συνεργαστούν που να βασίζονται και σε μια στρατηγική σοφά προετοιμασμένη με κατάλληλη αναρχίστρωση. Ακριβώς η νέα αυτή μορφή ενεργειών απαιτεί γενικές σφαιρικές απαντήσεις ε, και όλα αυτά έχουν σχέση με τα διπλωματικά, τα, οικονομικά, την ενημέρωση και το στρατιωτική πτυχή βέβαια. Στην Ουκρανία οι ενέργειες αυτές βλέπουμε ότι θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές η με την άλλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από από χώρες ακριβώς και σε εθνικό επίπεδο. Και στο Νότο βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει κρίση που, που είναι από την Αφρική, Βόρεια, την Περσαχάρια και βλέπουμε ότι μόνο μια γενική σφαιρική προσέγγιση θα μπορούσε τουλάχιστον να περιορίσει, να ελέγξει. Και για αυτή τη σφαιρική αντιμετώπιση θα πρέπει να δούμε τη Σομαλία που είναι κλασική περίπτωση. Τη βλέπουμε, παρατηρούμε ότι η σημαντικότητα των προσπαθειών ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, στην Αφρικανική Ένωση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, βλέπουμε ότι έτσι μειώθηκε και φαινόμενα πειρατείας ε, στις ακτές, αλλά βλέπουμε ότι κάπως περισσότερο ελέγχουμε την κατάσταση και σε ένα τομέα που έχει αμεσότερη σχέση με ε, στρατιωτικές μας δυνάμεις ή ε, αν ε, η ισχύση δυτική που υπερισχύαμε ακριβώ που εκεί βασιζόμαστε στις χώρες της, του ΝΑΤΟ εδώ και αρκετές δεκαετίες γιατί αλλάζουν όμως τα πράγματα. Βλέπουμε ότι εδώ και εκεί αναπτύσσεται στρατιωτική ισχύς ε, και τεχνολογική με αποδοτική. Γιατί δεν κοστίζει πια αυτή η τεχνολογία. Και άρα λοιπόν και οι αντίπαλοι μας ε, ε, γίνονται ισχυροί πια και υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι για τις στρατιωτικές μας δυνάμεις. Κοινή πρόκληση λοιπόν που συνόψα μόλις οι δύο αυτές οργανώσεις, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να έχουν μια κοινή, ένα κοινό όραμα. Και ε, ακριβώς την Επιτροπή αυτή η αλλαγής ε, ε, υποστήριξα ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει και να βασιστούμε στις προοπτικές, στην ανάλυση των προοπτικών για το μέλλον, τις δυνατότητες συνεργασίας και τα σχετικά έγραφα αυτά, οι μελέτες αυτές έχουν σημασία το μέλλον πολιτικά, ανθρώπινα, όσον αφορά τις τεχνολογίες σίγουρα, οικονομικά, με το περιβάλλον, όλα αυτά τα πράγματα να δούμε τι τα προκαλούν, ποιοι είναι οι παραγόντες αστάθειας, σίγουρα υπάρχουν και να δούμε και να βγάλουμε τις συμπεράσματα ακριβώ τι γίνεται σχετικά με τη στρατηγική μας και τη στρατηγική μας ικανότητα. Θα πρέπει στο μέλλον να δούμε πολιτικά πώς θα πού πρέπει να στραφούμε Όλα αυτά προετοιμάζονται βέβαια για ένα νέο κύκλο προετοιμασίας, ε, μια διαδικασία στατηρικού σχεδιασμού και θα έχουμε ένα νέο άξονα σημαντικό για τους δυο μας να προετοιμάσουμε μαζί το τι μπορούμε να κάνουμε, αυτά που θα απαιτηθούν, που θα χρειαστούμε αύριο. Θα συνεχίσω αγγλικά τώρα. Με δεδομένες τις προκλήσεις αυτές, Πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι να ανταποκριθούμε στρατιωτικά, να προωθήσουμε την ε, διαλειτουργική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα σε εκτυπήματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες επιχειρησιακές προκλήσεις. Απαιτείται προς τούτο ετοιμότητα και εκπαίδευση με βάση θεσμοθετημένες διαδικασίες χάρη και σε μια παράδοση διαβδουρικότητας δύο δεκαετιών. Στο Σικάγο πριν από δύο χρόνια έλαβαμε πρωτοβουλίες χάρη στις οποίες είμαστε πλέον σε θέση να συγχρονίσουμε εθνικές με ανατολικές ασκήσεις συμπεριλαμβανώντας και τους εταίρους στην Ανατολή. Έτσι, πλέον ασκήσεις με μεγάλη συχνότητα, μέρα παραμέρα σχεδόν, κατά το οποίο καλύπτει πλέον και την Ανατολική Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμπεριλαμβάνουν την προετοιμασία για υψηλού επίπεδου στρατηγικές ασκήσεις, Έχουμε, μάλιστα μια μεγάλη τέτοια άσκηση το 2015 με συμμετοχή Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας όπου πάνω από 25.000 στρατιωτικοί θα λάβουν μέρος. Αυτές οι ασκήσεις στον, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα και στον κυβερνοχώρο θα συμπεριλάβουν για πρώτη φορά τις χώρες ε, Βίσεγκραντ. Είναι μια μάλιστα άσκηση πιστοποίησης η οποία θα προσταθεί στην μεγαλύτερη άσκηση. Πρόκειται μια μεγάλη ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Όμως, είναι αλήθεια και το υπενθυμίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ετοιμότητά μα Αυτό απαιτεί επενδύσει στην εκπαίδευση και σε ασκήσει. Πρέπει να σταματήσουν οι μειώσει των αμυντικών προπολισμών. Αυτό το έχουμε τονίσει. Το τόνισαν στην Ουαλία και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το τόνισαν μάλιστα και σε Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Οι σύμμαχοι λοιπόν δεσμεύθηκαν να δαπανίσουν 2% του έπτους 20% του οποίου θα πάει σε επενδύσεις, σε έρευνα και τεχνολογία. Οι δαπάνε αυτές πρέπει να επενδυθούν με τρόπο έξυπνο, συνεκτικό, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός του ΝΑΤΟ. Ο σχεδιασμό ε, για το μέλλον είναι πολύπλοκη διαδικασία. Το ΝΑΤΟ έχει τις δικές του διαδικασίες, η ΚΕΠΑ έχει τις δικές της διαδικασίες. Το ΝΑΤΟ καθορίζει απαιτήσει, το πόσο θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτάται από μια ανάλυση μειονεκτημάτων, από δημιουργία βάσεων δεδομένων και τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Και οι δύο πάντω διαδικασίε, έχουν διαφορετική περιοδικότητα, όμως δεν βλέπω γιατί να μην προσπαθήσουμε πραγματικά να εξεύρουμε δυνατότητες συγχρονισμού, για να μην πω εναρμόνιση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την συμπληρωματικότητα των δύο διαδικασιών. Το ΝΑΤΟ Μπορεί αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη δική μα ανάλυση στο ΝΑΤΟ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την φιλόδοξη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013 να δίνουμε τη συνεργασία μας στους δορυφόρους, τα μη επιδρομένα οχήματα και στον κυβερνοχώρο. Ο στόχο είναι να εξασφαλίσουμε ικανότητε και να κλείσουμε τα κενά που υπάρχουν τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι και η ικανή απάντηση στο διαρκέ ερώτημα της κατανομής των βαρών. Προτιμώ κατανομή καθηκόντων και ευθυνών παρά βαρών. Είναι παλιό το ερώτημα. Είναι θέμα στο οποίο επιμένουν πάρα πολλοί οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Αυτά όλα σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΝΑΤΟ πρέπει να συνομιλούν, να ανταλλάσσουν απόψει και α πούμε στον ηλεκτρονικό χώρο. Η ομάδα εργασία με τον κυβερνοχώρο συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, α πούμε την περσμένη εβδομάδα, το σχετικό επιτελείο συμμετείχε στη μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση στον κυβερνοχώρο του ΝΑΤΟ. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας αντίλεξε πληροφορίες και συμμετείχε σε συσκέψεις όσον αφορά τις ηλεκτρονικές δυνατότητες στο Τάλιν της Εστονίας. Ο συντονισμός λοιπόν είναι παρόν, είναι εξαιρετικά επικοδομητικός μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ε, και της αντίστοιχη δομή των ΝΑΤΟ. Έχουμε την πρωτοβουλία για την έξυπνη άμυνα. Οι προσπάθειες, επαναλαμβάνω, είναι συμπληρωματικές. Είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό και είμαι σίγουρος ότι μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτήν την πως συντονισμού. Το αν οι ικανότητε θα αναπτυχθούν υπό τον ΝΑΤΟ ή υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση οι δομέ αυτέ πρέπει να είναι κοινέ και να είναι στη διάθεση και του ενό και του άλλου οργανισμού. Οποιοδήποτε και οπουδήποτε τη χρειαστεί προ το όφελο και των δύο οργανισμών. Συνεπώ, στον τομέα τη καινοτομία βρίσκω πολύ ενδιαφέρον να έργο στο οποίο είχα συμμετάσχει πριν από μερικά χρόνια. Είναι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφορών, πρωτοβουλία τεσσάρων χωρών, συντονισμού στον τομέα των αερομεταφορών. Πηγαίνει πολύ καλά και έχει ωφελήσει και το ΝΑΤΟ και τις εθνικές επιχειρήσεις. Και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι και άλλες χώρες, μαζί με τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, συμμετέχουν στην προσπάθεια. Η Ισπανία είναι ήδη μέσα, το εξετάζει το ενδεχόμενο και η Ιταλία. Πρόκειται για μια πολύ έξυπνη θα έλεγα προσέγγιση στα προβλήματά μα. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην Ευρώπη, αερομεταφορική ικανότητα. Πρέπει λοιπόν να μοιραστούμε αυτά που έχουμε, να τα συγκεράσουμε καλύτερα και να κάνουμε οικονομίες επενδύσει. Υπάρχουν όμω και άλλα παραδείγματα για να παραμείνω στις αερομεταφορές. Ο αντίπαλος το σκάφος α Α400M ήδη είναι έτοιμο με την υποστήριξη του ΟΚΑΡ και του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μια ουσιαστική συνεργασία. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει θέση στο έργο του ΝΑΤΟ να αναπτύξει τις αμυντικές μας δυνατότητες και αυτό τονίστηκε και στην Ουαλία. Η μορφωσή του ΝΑΤΟ θα ωφελήσει την βιομηχανία και στις διόχθες του Ατλαντικού. είναι η δίκαιη επιστροφή για όλους. Τις επόμενες δεκαετίες θα έχουμε στολό iWalks, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε τόσες πολλές περιπτώσεις. Ο στόλος αυτός πρέπει βεβαίως να ανανεωθεί. Εμεί θα προβούμε σε επιχειρησιακή ανάλυση για ένα πολύ πολύπλοκο σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να γίνει και αιχμή του δόρατος της ε, αμυντική μα συνεργασία στον τομέα τη βιομηχανία. Τα συστήματα δική και ελέγχου θα βρεθούν επιπλέον, ε, καθώς και η συνεργασία στον κυβερνοχώρο. Όλες οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη περιφερειακή αυτή προετοιμασία είναι για να μπορέσουν να μπορούν να αντιδρούν άμεσα οι δυνάμεις μας. Και στην Ουαλία είδαμε την αντίδραση και το σχέδιο για αυτό για να μπορούμε άμεσα ε, να ανταποκρινόμαστε από την πρόκληση στα σύνορα και το ΝΑΤΟ έχει μια δύναμη που να μπορεί εύκολα την ZTF να μπορεί σε λίγες μέρες να είναι επιτόπους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε ακόμα να προσδιορίσουμε τις λεπτομέρειες αλλά σίγουρα θα αποτελεί ε, σημαντικό βήμα και απαιτεί σημαντικές προσπάθειες. Θα είναι να δοκιμή αλληλεγγύης αλλά επίσης θα βασίζεται και στα κεκτημένα για τις ε, άμεσες δυνάμεις κρούσης άμεσης ε, εδώ και εκεί ε, και αμερικανικής πλευράς και Ευρωπαϊκή πλευρά. Έστω και αν αυτέ οι οι δυνάμεις αυτές ε, δεν πάνε για τι ίδιε αποστολέ. σίγουρα όμω είναι συμπληρωματικέ και θα πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται μόνιμα και σταθερά. Επίσης για την αυτιλιακή ασφάλεια αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το θέμα σημαντικό είναι, καλύπτει πολλά σημεία και στο ΝΑΤΟ ακριβώς που να μπορεί να είναι επιχειρησιακά αποτελεσματικό και θα πρέπει να όσο γίνεται περισσότερο οι να είναι συμπληρωματικές ε, και να υπάρχει ένα κοινό στρατηγείο ναυτικού σχεδιασμού και θα ήθελα να επιμείνω επίσης σε κάτι άλλο. Δύο κοινού ενδιαφέροντος τομείς, σημαντικούς τρομερά για τη διαχείριση κρίσεων και άλλων απειλών όπως βλέπουμε σήμερα, να μπορούμε πριν να προλαβαίνουμε την κρίση και την επικοινωνιακή στρατηγική και θα θυμηθούμε τις κρίσεις είτε την Αραβική Άνοιξη, την Ουκρανία είτε ε, της ε, κρίσης στη Συρία και στο Ιράκ ε, θα πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να μπορούμε να τα προλαβαίνουμε. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το να μπορούμε πριν να ξεσπάσει η κρίση να προλαβαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον ΝΑΤΟ είναι σημαντικά. Είναι και τρομερή δυνατότητα συνεργασίας πολιτική και στρατιωτική. Επίσης ε, μια στρατηγική πραγματικά ενεργό δράση πάνω σε κρίσεις στην Ουκρανία ας πούμε που βλέπουμε συνεχώς ε, οι Ρώσοι ότι είναι πόσο καλά ενοργανωμένοι στο Ιράκ και που ακριβώς ε, είναι χρησιμοποιούν εκεί οι ε, φανατικοί τις δυνατότητες επικοινωνίας τους. Εδώ θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και από τις δύο πλευρές και θα αποτελούσε αυτό ένα σημαντικό βήμα. Κάτι ακόμα. Ολοκληρώνοντας με μια ρεαλιστική επικοδομητική αντιμετώπιση της διαχείρισης των κρίσεων, τις δυνατότητες που έχουμε, ε, ασκήσεις των δυνάμειών μας, ε, μια επικοινωνική ε, μια επικοινωνία στρατηγική. Έτσι οι χώρες μας ε, θα έχουμε δυνατότητες να ενισχύσουμε αυτή την πνευματικότητα. Κοινή προσπάθεια είτε στο κέντρο Αφρική, στα Βαλκάνια και στο Αφγανιστάν ε, και στη Μεσόγειο. Αυτό αποτελούν λόγους κατάλληλους για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο και επίσης να επενδύσουμε και πάλι στην άμυνα στις ευρωπαϊκές χώρες και στην στη σκέψη κορυφή αλλά και στη, στην σύσκεψη του ΝΑΤΟ να ενισχύσουμε τις δυνατότητες μας στρατιωτικέ μα, και να είναι αξιόπιστε, στα πλαίσια τη όλης οργάνωση και στο ΝΑΤΟ βέβαια. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι κύριε Πρόεδρε. Το Γενικό Στρατηγείο ακριβώς προσπαθεί να ενισχύσει αυτή τη διάφανη ανοιχτή συναντική συνεργασία που να σέβεται ταυτόχρονα και την αυτονομία και την θεσμική ανεξαρτησία των οργάνων σας. Σας ευχαριστώ και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε κάθε ερώτηση. Ευχαριστώ στρατηγέ μου, λέει Πρόεδρος. παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, στρατηγέ. Από την παρουσία σας βλέπω ότι η κύρια μεταμόρφωση στο ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια αφορά την ένταξη των νέων κρατών από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Χώρες οι οποίες για δεκαετίες εκδήλωναν εχθρότητα απέναντι στον ΝΑΤΟ. Ίσως αυτές οι αντιλήψεις να παραμένουν για ορισμένους. Εγώ στην Τσεχία σε σημαντικά πολιτικά κόμματα τέτοιου είδου εχθρότητα και κατάλοιπά τη. Επί παραδείγματι στο σχεδιασμό για την εξωτερική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχίας που είναι σημαντικό κόμμα στο κοινοβούλιο της χώρας ε, υπάρχει ο σχεδιασμός για την αποχώρηση από τον ΝΑΤΟ. Και υπάρχει αν θυμάστε και η ε, πρόθεση της κυβέρνησης ε, να υπογράψει συμφωνία για την εγκατάσταση δορυφόρων στη χώρα, μάλλον ραντάρ στη χώρα, που δεν ενέκρινε το κοινοβούλιο. Πώς μπορείτε λοιπόν να έχετε μια ενιαία προσέγγιση προς τα μέλη του ΝΑΤΟ στο σύνολό τους ή μήπως τελικά έχετε διαφορετικά, διαφορετική προσέγγιση και ανάλογα με την ημερομηνία προσχώρησης της κάθε χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσω όμως ε, τις ερωτήσεις μου, έχω να ρωτήσω το εξής, γιατί μπορεί να έχω παρεξηγήσει κάτι. Εσείς είσαστε ο διοικητής ACT του Norfolk, έτσι. Καλώς. Ωραία. Αυτό το κέντρο λοιπόν από ό,τι γνωρίζω αφορά δύο οργανώσεις στο Στάβανκερ της ε, Νορβηγίας και το Πίτκος της Πολωνίας. Έτσι, δύο μονάδες το ΣΥΠΗΝ που, που δρούν στην Ευρώπη. Ωραία, άμα το έχω καταλάβει αυτό θα είναι και πιο εύκολο να δείτε πώς θα τις ερωτήσεις μου. Γιατί δεν το αναφέρατε. Α, ναι, και μία στην Πορτογαλία πολύ καλά. Μιλήσατε αρκετά εκταμένα για την ανάγκη να διατυπωθούν κοινά συμπεράσματα για τις αλλαγές στη στρατιωτική κατάσταση και γενικά τη συμμαχία. Πριν από δύο μέρες ήμουν στον Πίτκος, τυχαία ξέρετε, στο κέντρο αυτό που συστήθηκε πριν από δέκα χρόνια. Ένα κέντρο για το οποίο είναι υπερήφανη, τα Μάλα, η Πολωνία και το οποίο υπηρετεί ψηλά λειτουργήματα στη χώρα. Είναι πολύ σύγχρονο. Πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από το δυναμικό κατάρτισης που υπάρχει εκεί. Έχω όμως την εξής ερώτηση. Αυτά τα κέντρα που έχουν ιδρυθεί μέχρι τώρα εστιάζονται στην εξασφάλιση της κοινή διοίκηση για τις επιχειρήσεις ΙΣΑΦ, οι οποίες όμως τώρα εκπνέουν καθώς αλλάζει το ρόλο του στο Αφγανιστάν τον ΝΑΤΟ στον το χρόνο. Ερωτώ λοιπόν. Από εδώ και μπρο αυτά τα κέντρα, τα τόσο σύγχρονα ευρωπαϊκά κέντρα που έχουν πάνω από 20 από, έχουν προσωπικό προερχόμενο από 20 και πάνω χώρες τι θα κάνουν από εδώ και μπρο. ξέρετε είναι κάπως αβέβαιο το μέλλον αυτό είναι το ένα ζήτημα το δε άλλο σχετίζεται με συζητήσεις που πραγματοποιούμε στην Επιτροπή μας και αφορούν τις σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες οι οποίες θέλουν φερειπή να ανακηρύξουν την ανεξαρτησία τους όπου φαντάζομαι πως δεν χρησιμοποιείται τα κέντρα αυτά για τέτοιου είδου αλλαγέ σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή θα ρωτούσα πόσους έχουμε από τη Γεωργία εκεί. Έναν. Από την Ουκρανία. Άλλον ένα. Που επίσης προτιμούσε να είναι εκεί πέρα από ότι ε, οπουδήποτε αλλού, ας το πούμε έτσι. Και έχω την εξή ερώτηση. Έχουμε τόσα, τόσο καλά μέσα, προσωπικό, καταρτισμένο και ικανό δεν θα έπρεπε να ενισχύσουμε την κλίμακα της αξιοποίησης των κέντρων αυτών για την κατάρτιση των στρατιωτικών των χωρών εκείνων που χρειάζονται καλό στρατιωτικό προσωπικό για να μπορεί να υπερασπιστεί την ασφαλεία τους. Δηλαδή όταν, εάν δούμε ότι μπορεί να χρειάζονται βοήθεια, μπορούμε να τους μοιράζουμε Αλεξίς Φεραγγιλέκα, αλλά πραγματικά χρειάζονται κατάρτιση. Ο κύριος Βανόρτεν έχει το λόγο. Uh, <coughs> ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Θεωρείτε ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι πολιτικού χαρακτήρα, ό,τι όνομα ή διαμόρφωση και αν έχει. Ε, και όχι στρατιωτική. Και δεν χρειάζεται να περιπλέκονται οι σχέσεις μας με τον ΝΑΤΟ. Γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος ούτε καν πόρη για επικάλυψη και σπατάλη δραστηριοτήτων. Μιλήσατε για βιομηχανικά έργα. Κανένα από αυτά όμως, για να είναι σαφές, δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έργα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων υπό την αιγίδα της ΟΚΤΑ ή άλλων οργανισμών, αλλά όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ρωτήσω από τη γενική θεώρηση εκ του μηδενός για την ρύθμιση, εάν θεωρήσατε ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει ενσωμάτωση ή ανάγκη ενσωμάτωσης κάποιων ευρωπαϊκών οργανισμών στο ΝΑΤΟ. Η Στρατιωτική Επιτροπή, παραδείγματι, θα μπορούσε να διαρθρωθεί κατά τρόπον τέτοιο που όταν υπάρχουν δραστηριότητε στις οποίες θα έπρεπε να ηγηθεί ε, μια ευρωπαϊκή χώρα θα έπρεπε να σε θέσει να λαμβάνει η Στρατιωτική Επιτροπή τέτοιες ε, αποφάσεις. Γι' αυτό δεν υπάρχουν προηγούμενα από ό,τι γνωρίζω. Και επίση για να συνεχίσω, ξέρουμε ότι η Γαλλία έχει πιστεύω τις ευθύνες της για την δημιουργία μιας χωριστής κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Και πρέπει η Γαλλία από τη μοναδική της θέση να αναγνωρίσει το λάθος και να δώσει νέα πνοή σε μια φρέσκια προσέγγιση. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα και δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά όπως παίζουμε. Εσείς από τη θέση σας καταλαβαίνω βεβαίως ότι οφείλετε να υπηρετήσετε τουλάχιστον ε, στα λόγια την ε, κοινή Επιτροπή Ασφαλείας και Άμυνας και αυτή είναι η δουλειά σας αλλά συμπληρωματικότητα δεν έπρεπε να υπάρχει ανάγκη να αναζητούμε στη τελευταία ανάλυση τα ίδια κράτη είναι διαλειτουργικότητα η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων έπρεπε να είναι δεδομένη και δι διαλειτουργικότητα μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αλούζη. Η κυρία Λέζινγκ χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να διατυπώσω κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις για θέματα που διάβασα στον τύπο ή από άλλες πηγές που μπόρεσα να αντλήσω πληροφορίες που αποδεικνύονται τελικά αντιφατικές. Η μία ερώτηση έχει να κάνει με τις ε, δυνάμεις ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ, όπου λέτε ότι θέλετε 4 με 5 χιλιάδες ε, στρατιώτες να περιληφθούν. Με παρακολουθείτε ενώ ο Hans Luther Domröse, στρατηγός Γερμανός του ΝΑΤΟ, ανέβασε τον αριθμό αυτό στις 7.000 στρατιώτες. Ερωτώ λοιπόν, είναι σωστό αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Ντομρόζε ή όχι, εσείς ε, για τα μεγέθη αυτά τι έχετε να πείτε. Και επίση ο κύριος Ντομρόζε μίλησε επίσης για μεγάλες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ μέχρι 40.000 ανδρών άσκηση που θα αναπτυσσόταν πολύ κοντά στα ρωσικά σύνορα. Μπορείτε αυτό να το επιβεβαιώσετε. Και κάτι ακόμη για το Αφγανιστάν. Οι New York Times έχουν ε, ε δημοσιεύσει ότι στο Αφγανιστάν το ΝΑΤΟ θα έχει 14.000 στρατιώτες. Ισχύει αυτό και αν ναι, από ποια κράτη και σε ποια αναλογία θα προέρχονται οι στρατιώτες αυτοί. Στη Reuters διαβάζω 27 Νοεμβρίου ότι ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έδωσε άδεια για αποστολή Αμερικανών στρατιωτικών για την ανάληψη και επιθετικής δράσης και κυρίως την ε, ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση των Ταλιμπάν. Αυτό είναι αντίθετο με αρχικές αναφορές ότι θα, έπαυ, θα έπαβε στα τέλη του 2014 η στρατιωτική εμπλοκή των Αμερικανών. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, να μου δώσετε κάποια απάντηση. Ευχαριστώ. θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Κλώτ Φρανς Αγνώ, την επικεφαλής εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας και η οποία θα μιλήσει ευθύ αμέσως. Αλλά προηγουμένως ο κ. Φαντουλίτσα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε και αυτά που επιτελέσατε σαν επικεφαλής ακριβώς ε, του μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ από το 2012. Πεστε μου σας παρακαλώ, τα μέτρα που έλαβε το ΝΑΤΟ ή που θα λάβει το ΝΑΤΟ κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη για να απαντήσει στις προκλήσεις της Ρωσίας στη θάλασσα της Βαλτικής, στην Μαύρη Θάλασσα και αλλού, σε άλλες ε, περιοχές της Ευρώπης και του Ατλαντικού. Στρατηγέ μου, πέστε μου σας παρακαλώ. Το ΝΑΤΟ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τι καινούργια τμήματα θα έχει για να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις και για την άμυνα την ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ, στρατιέ. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ε, κοινοβουλευτικής συνόδου, ο Γερικός Αμαθέας, ο κύριος Στόλτενμπεργκ, μίλησε για την δημιουργία δυνατοτήτων δυνατοτήτων και υποπίλητης ε, υπέρ των ανατολικών γειτόνων και δι της Ουκρανίας. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κατάλληλος των μιλητών έχει κλείσει, οπότε ο λόγος των στρατηγικών παλαμέρων και τα κυρία Αρνό. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας. Ήταν εξαιρετικά εύστοχε οι ερωτήσεις. Όμως ε, να τονίσω ευθύ αμέσως ότι σε καθημερινή βάση λειτουργούμε με τρόπο που αποδεικνύει ότι όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ για μας είναι σημαντικά τα οποία πρόσφατα στην Αλβανία, στην Κροατία και βλέπω παντού εξαιρετικά αποτελέσματα, εξαιρετική προσήλωση στόχους του ΝΑΤΟ. Ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφίας. Όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι παρόντα, συμμετέχουν, κατανοούν τις ευαισθησίες των προκλήσεων και η δική μου ανάγνωση της Ουαλίας ήταν ακριβώς απόδειξη της προσήλωσης αρχικών κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών. Πρέπει να πω ότι με γέμισε ενθουσιασμό η προσήλωση όλων και των 28 αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, είναι αλήθεια ότι Είμαι διοικητή τριών ουσιαστικά διοικήσεων στην Ευρώπη και ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί έχω την ευκαιρία να τονίσω την αξία όλων των ανθρώπων, των στρατιωτικών οι οποίοι υποστηρίζουν την μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ. Ο κ. Στάβενγκερ, ο οποίο είναι επικεφαλή του Joint Warfare Center, τον Bill Koch, ο οποίο είναι υπεύθυνο προετοιμασία και ο οποίο βρε τα μέγιστα στην προετοιμασία της αποστολή στο Αφγανιστάν. Ε, ε, προετοιμασία πολλές ε, ασκήσεις επίσης. Στην Λισαβόνα επίσης έχουμε το κοινό κέντρο αναλύσεων. Πρόκειται για τρεις πυλώνες της αλλαγής του ΝΑΤΟ. Κλειδί για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι ας πούμε στον τομέα της διαλειτουργικότητας γίνεται πάρα πολύ δουλειά. στο μέλλον θα είμαστε όλο και πιο προετοιμασμένοι χάρη σε γυμνάσια γιατί έχουμε τις γνώσεις, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε την πλήρη υποστήριξη της Πολωνίας και άλλων χωρών φυσικά. Συνεπώς είμαι πολύ πεπισμένος ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις διοικήσεις, αυτά τα αρχηγεία για να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την διαλειτουργικότητα. Όπως ξέρετε Αυτό είναι ένα από τους βασικούς στόχους μου πρώτα που ανέλαβα. Και ξαναθυμίζω ότι ο στόχος ε, η πρωτοβουλία Key Force Initiative θα συνεχιστεί. Υποστηρίζουμε επίση του εταίρου μα μέσω αυτού που ονομάζεται πλατφόρμα διαλειτουργικότητα για του εταίρου. Και τονίζουμε τη δημιουργία αμυντικών δυνατοτήτων. Αυτό το είπαν και οι αρχικοί κρατών κυβερνήσεων στην Ουαλία. Είναι βασική προτεραιότητα, προτεραιότητα κλειδί για τη Γεωργία σίγουρα, για την Ιορδανία, τη Μολδαβία και ίσως αν χρειαστεί ε, και στο Ιράκ η Ιρακινή κυβέρνηση ρώτησε αν μπορεί να τη βοηθήσει στο ΝΑΤΟ και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει η Γεωργία σίγουρα πάνω και η Ουκρανία η Ουκρανία ε, εδώ και χρόνια είναι εταίρος του ΝΑΤΟ ήταν εταίρος όχι μέλος βεβαίως το τονίζω αυτό γιατί πολλοί ρωτάνε τι κάνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία το ΝΑΤΟ έχει εξαιρετική συνεργασία με την Ουκρανία η Ουκρανία συμμετέχει σε επιχειρήσεις μας μεταξύ αυτών και στο Αφγανιστάν. Η αποστολή αυτή αξιοποιεί 12.500 στρατιωτικούς με τη συμμετοχή και εταίρων. Πρόκειται για μια αποστολή η οποία έχει αφιερωθεί στην περιοχή συμβουλών και εκπαίδευσης το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούν εκεί με αυτά που λέμε παράγοντες καταλητικούς παράγοντες κλειδιακοί enablers αυτά τα οποία δεν έχουν ακριβώς οι Αφγανοί αεροπορική υποστήριξη κεντρικές υπηρεσίες μεταφορές ιατρικού χαρακτήρα Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ του Αφγανού, ε, οι οποίοι μαθαίνουν, βελτιώνονται κάθε μέρα Σίγουρα εκεί είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Όσον αφορά την εντολή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και του κανόνε εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι δικέ του δυνάμει, ακούσατε τον πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίο δήλωσε ότι θα δώσει πιο συγκεκριμένου κανόνε εμπλοκή στι δυνάμει του για να μπορούν να αυτοπροστατευθούν και αφού σου σε στα καθήκοντά του στην υποστήριξη των Αφγανών. Πολύ σημαντική απόφαση για την οποία εκφράζω την ικανοποίησή μου. Τονίζω ότι στην επόμενη αποστολή που ξεκινάει 1η Ιανουαρίου του 2015, Resolute Support, το προσωπικό δεν θα έχει επιθετική αποστολή παρά να βοηθήσει τους Αφγανούς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και σήμερα. Ξέρουμε ότι θα ενταθεί η πίεση από τους Ταλιμπάν, γιατί αυτοί γνωρίζουν ότι συρρυκνούνται η παρουσία του ΝΑΤΟ. Πάντω οι δυνάμει ασφαλεία του Αφγανιστάν πλέον είναι σε θέση με τη βοήθειά μα και την υποστήριξή μα να αναλάβουν τον ρόλο τη υπεράσπιση τη χώρα. Όσον αφορά την τιμότητα τη Task τη δεμής ακούσατε διάφορα νούμερα. Το χερσαίο τμήμα θα αποτελείται από 4.000 με 5.000 άνδρες, είναι σύντομα έτοιμοι, αλλά υπάρχει και ο αεροπορικό κλάδο και βέβαια στο κέντρο ελέγχου και διοίκηση. Όπω είπα, στην ξέρα θα έχουμε περίπου 5.000 άνδρες. Το σύνολο μπορεί να φτάσει στους 10.000 μαζί με την αεροπορική συνιστόσα και τη θαλάσσια συνιστόσα. Βασικά μιλάμε για μια ταξιαρχία. Ένα σώμα ταξιαρχίας γύρω στις 5.000 ε, και γυναίκες. Τώρα, για και ΚΕΠΑ, τον ΝΑΤΟ, τις επικαλύψεις, άκουσα πολλές ερωτήσεις. Ε, κατανοώ από πολιτικές όψεως τι δηλώσει αυτέ Δεν θα το σχολιάσω αυτό από την παρούσα θέση μου, ούτε έχω διηγήσει τη χώρα μου. Εγώ είμαι ανοίγω στο ΝΑΤΟ, κάνω πράγματα για τις 28 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει εξασφαλίσει την ειρήνη για 28 χώρες εδώ και δεκαετίες, για 65 χρόνια συγκεκριμένα. Η Γαλλία επανήλθε στο στερεωτικό σκέλος, ο χάρηκε για αυτή την εξέλιξη και δεν ήξερα βεβαίω τώρα ότι θα γινόμουν επικεφαλή ε, ενός μιας ανατολική διοίκησης. Όσον αφορά τη δική σα αποστολή, εσείς και άλλοι βεβαίω τονίζουν τον κίνδυνο επικάλυψη. Το πρόβλημα δεν είναι η επικάλυψη σήμερα. Το θέμα είναι να καλύψουμε τις ελλείψεις μας και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το αν αυτό που κάνω ε, ανήκει αν θέλετε στη Γαλλία ή στο ΝΑΤΟ δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι πώς θα βελτιώσουμε τις δυνατότητες μας, τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών χωρών. Και τα 28 οι μελη καλούνται να συνεισφέρουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει επικάλυψη. Και πάση περιπτώσει, αν υπήρχε, θα το λύναμε το πρόβλημα. Όμως το βασικό είναι η ελλείψη που έχουμε στις ικανότητες μας, στις αμυντικές μας δυνατότητες. Γι' αυτό και εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρωτοβουλία στο επίπεδο των δορυφόρων, των μη παντανομένων αεροσκαφών, των, του ενεργείου ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής. Και για να απαντήσω και την άλλη ερώτηση, θα βλέπω τη σύσταση, τη σύνθεση της Στρατηγικής Επιτροπής. Πρέπει να σας πω ότι η συντηρητική πλειονότητα των μελών, και το γνωρίζετε, με μέλη και τη αντίστοιχη επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό αυτό. Η διαπολιτική οπτική. Υπάρχουν κατά τα άλλα αποστολέ που καλύτερα τις εκτελεί το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν άλλες αποστολέ όπου ίσως το ΝΑΤΟ δεν έχει τόσο θέση. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πιο αποτελεσματική. Και εκεί χρειάζεται προετοιμασία. Να λοιπόν που υπάρχει συμπληρωματικότητα, όχι επικαλύψεις. Και να πως ε, διευρύνεται το πεδίο και το αντικείμενο των αποστολών μας. Γι' αυτό θα το ξαναπώ, η διαλειτουργικότητα είναι μεγάλη σημασία, η εκπαίδευση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση. Φυσικά θα κοιτάξουμε να αποφύγουμε επικαλύψεις, και μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με άλλου οργανισμού. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητέ μα, Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε με διαφορετικά πρότυπα γιατί εν τέλει οι ίδιοι οι ίδιε γυναίκες θα ριχθούν στο πεδίο τη μαχη αν χρειαστεί και εκεί θα χρειαστεί η διαλειτουργικότητα. Νομίζω δεν απήντησα στο θέμα που αφορά τη Ρωσία και τις προκλήσεις. Νομίζω γνωρίζετε ότι το ΝΑΤΟ έχει παράσχει διαβεβαιώσεις με συγκεκριμένα μέτρα μετά από αυτά που έγινε στην Ουκρανία. Για να διασφαλίσουμε ότι αν χρειαστεί θα ενισχύσουμε την παρουσία μας και τη θέση μας ήδη οθετήσαμε μια δυναμική στάση δείξαμε ότι το ΝΑΤΟ είναι εδώ Ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε και προετοιμάζουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να ελοποιήσει τη βασική του αποστολή. Συλλογική άμυνα. Και αυτό που κάνουμε σήμερα το κάνουμε με τις γνωστές ασκήσεις στα γυμνάσια. Όπως είπα, έχουμε μια διαφορετική άσκηση σχεδόν κάθε δύο μέρες. Τώρα θα χρειαστούν νέες διοικήσεις για να αντιμετωπίσουν τη νέα συγκυρία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ακόμη συζητούμε. Όπως ξέρετε η μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ συνεχίζεται, ανεδιαρθρώνεται, το θέμα είναι να γίνει πιο αποτελεσματικό, όπως και η δομή διοίκησής του. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι προς το παρόν <laughs> βολευτείτε με αυτά που έχετε. Πάντως κάποια στιγμή θα ε, ε, Ξέρετε ότι έχουμε μια βασική διοικητική δομή και από εκεί πέρα έχουμε τις δυνάμεις. Πρέπει να συνδυάσουμε τις εθνικές συνεισφορές με την κεντρική δομή του ΝΑΤΟ που όπως είπα δεν μπορεί να μεγαλώσει άλλο. Το ΝΑΤΟ λοιπόν συνεχίζει ε, να αλλάζει αλλάζει διαρκώς σε αρτήση των εκάστοτε προτεραιοτήτων. Αυτά νομίζω. Α, και άλλη μια ερώτηση που νομίζω δεν απήντησα. Χθε ε, για τη Γεωργία ετέθη το σχετικό ερώτημα. Ε, εδώ θέλω να τονίσω ότι πολλοί Υπουργοί, χωρίς να επισέλθουν σε λεπτομέρειες, είπαν ότι και εδώ, προκειμένου, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα των επικαλύψεων. Πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα και σίγουρα η γεωργία είναι προτεραιότητά μας. Στην προσπάθεια δηλαδή ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρα το είπαμε και χθε. Όπως άλλο το κάναμε και στο Αφγανιστάν. Πρόεδρος, ευχαριστώ στρατηγέ. Παρακαλώ παραμείνετε για, και την δεύτερη συνεδρία μας. Και τώρα να καλωσορίσω την κυρία Κλοντ Φρανς Αρνού, εκκλησιαστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Εκκλησίας Άμυνας. Η εντολή της τελειώνει τον Ιανουάριο του 2015, οπότε υπό μία έννοια είναι σχεδόν σε θέση να ανακεφαλαιώσει τα αποτελέσματα τη θητείας της. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει να συνεισφέρει πολλά από άλλη θέση. Παρακαλώ, κυρία, ενημερώστε μας για την κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και για την προσπάθεια δημιουργίας δυνατοτήτων στο πλαίσιο της ε, ΕΠΑ. Γνωρίζω, κυρία Μογκερίνη, σας επισκέφθηκε προσφάτως και συμμετέσχε στην συνεδρίαση της Επισπέδουσας Επιτροπής. Νομίζω ότι για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο. Οπότε, παρακαλώ κύριε Νου, ε, σας ακούμε. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ρυθμίσουμε το μικρόφωνο μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πρόκειται για μεγάλη τιμή και χαρά να έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας στο Ευρωπαϊκό και κατά τη διάρκεια της θητείας μου που λύγει βέβαια τον Ιανουάριο εποφεληθήκαμε εδώ από τη συνεργασία αυτή με την υπεπιτροπή σας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δόθηκε μια σημαντική όθηση σε αυτές τις εργασίες μας ε, για τις δυνατότητες, για τη βιομηχανική βάση και για την τεχνολογία άμυνας ε, και ασφάλειας στην Κίνη. Χαίρομαι που εδώ στο τέλος θητείας μου έρχομαι εδώ και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή ακριβώς ε, μετά από μια πολύ σημαντική φάση που παραμένει σημαντική μέχρι τον Ιούνιο ιδιαίτερες πολιτικές οθήσεις από το δεύτερο εξάμεινο και περισσότερο θα δούμε για την, ε, ε, το τι θα προκαλέσουν όλα αυτά σε υψηλότερο το επίπεδο μάλιστα και αυτή η αλληλεπίδραση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά με την Υπερεπιτροπή σας είναι κάτι το σημαντικό. Παίζεται ένα πολύ κεντρικό σημαντικό ρόλο, αρμοδιότητα και νομοθετική και προπολογισμού, ώστε όλες αυτές οι ιδέες που επικυρώθηκαν σε επίπεδο αρχηγών κρατών κυβερνήσεων να μπορέσουν να υλοποιηθούν νομοθετικά και οικονομικά στον προπολογισμό. Αυτές οι ενέργειες απαιτούνται περισσότερο από ποτέ. Και εδώ πώς έχει κατάσταση η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συνομβουλίου και για όλες τις εντολές υπήρξε μια βελτίωση. Πρώτα απ' όλα φιλόδοξα γιατί θέλαμε σε 4-10 προγράμματα να προχωρήσουμε. Δεν είναι ότι προσέχουμε μόνο αυτά τα τέσσερα προγράμματα. Πάντω από τη στιγμή που θα πετύχουν αυτά τα προγράμματα τι σημαίνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα και στην, ε, ε τον εφοδιασμό, τον αέριο εφοδιασμό, την ο, με τον στρατηγό Ζαμπον Παλωμέρο συζητήσαμε το 80% του αερίου φωδιασμού, τον εφοδιασμό επτήση θα γίνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο προσαρμός του Πενταγώνου είναι σαφής ότι θα πρέπει όμως ταυτόχρονα λένε να μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και ας πούμε για τη Λιβύη. Μην ε, υπολογίζετε σε εμά όπως συνήθως για το 80% της, ε, του εμπτήση ανεφοδιασμού. Αυτό λοιπόν, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα θα θέλατε να υποβάλλετε. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να υποφελθούμε όσο γίνεται από τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας τώρα, όπως στην Ιταλία. Νέα δυνατότητα σε σχέση με το παρελθόν. Βασίζεται στα Boeing και στο Ευρωπαϊκό Ιδρύμα για να δούμε ε, ανάλογα το με τις δυνατότητες εμπτής εφοδιασμού, να δούμε και τα είδη αεροσκαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και αυτό πειραματικά έτσι βλέπουμε, όχι δηλαδή σε στιγμή μάχης, βλέπουμε τις δυνατότητες που έχουν οι Ευρωπαίοι βάσει και αυτής της δυνατότητας της Ιταλικής. Αλλά το πιο φιλόδοξο σχέδιο ποιο είναι. Να έχουμε στόλο επιπλέον για, την, για τον επτήσιο εφοδιασμό το χρειαζόμαστε και διάφορες χώρες υπό την Ολλανδία εργάζονται για επιπλέον δυνατότητες ε, αεροσκαφών για που μπορούν να παίξουν πολλαπλούς ρόλους ας πούμε και για ιατρική, φροντίδα κλπ. Να δούμε λοιπόν και αυτή την, τον επτήσιο εφοδιασμό με την συνεργασία όσο γίνεται περισσότερο και με τη δυνατότητα του Ηνωμένου Βασιλείου ε, χάρη στη συμφωνία που έχει υπάρξει και από την πλευρά των Γάλλων με την πρόσφατη ε, συμφωνία για ε, την αγορά αεροσκαφών ε, για πολλαπλούς ρόλους ε, και μέσα από τη Ολλανδία θα περάσουμε τώρα με διαπραγματεύσεις με το τομέα της βιομηχανίας για να μπορούμε να επιλέξουμε το αεροσκάφος το επόμενο, το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες. Λέγεται το τηλεκατευθυνόμενο σύστημα πλοήγησης για μένα είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα. Τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο ωφέλιμα με τη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδείξουμε αυτό που απάντησε τον κύριο Βανόρντεν ο στρατηγός. Πώς μπορείτε να το αποκαλείτε αυτό σαν ε, υπερβολικό. Ναι. Εδώ λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, τις εργασίες. Ε, νομίζουμε ότι θα μπορούσαν να συγκλίνουν τα διάφορα στοιχεία και έτσι τα κράτη-μέλη, όπως το είπε και ο στρατηγός, αυτά είναι τα ίδια και μια μεριά την άλλη έχουν δυνατότητες τις οποίες θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ανάλογα με την πολιτική απόφαση. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση. Εμείς ε, πώς θα ωφεληθούμε στα πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα για την επόμενη γενιά αεροπλοήγησης τηλεκατευθυνόμενης ε, να είναι αυτή ασφαλής ε, κανονικά στο συνδυσμένο εναέριο χώρο. Και απαιτείται μια ρύθμιση κατάλληλη και θα πρέπει να το κάνει η Επιτροπή βασιζόμενη στα σχεδόν μέχρι τώρα και να έχουμε επίσης μια κατάλληλη τεχνολογική εξέλιξη που να μπορούσαν αυτά να ισχύσουν στον εναέριο αυτό χώρο και μια εργασία που γίνεται και στα πλαίσια ακριβώς του φορέα μας με με το Jeep Joint ε, Investment Programs όπως τα αποκαλούμε στα αγγλικά και επίσης δυνατότητες τρομερές ε, συνδυασμού και συνεργασίας ανάμεσα αυτά που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και στην εξέλιξη προς έναν νέο ε, ένα αέριο χώρο και με τις δυνατότητες τεχνολογικές για να μπορέσουν αυτά να ισχύσουν στον αέριο χώρο ακριβώς. Αρκετά πολλά στοιχεία τεχνολογικά, πολλές δυνατότητες μπορούν να ισχύσουν γιατί αποσκοπούν στην ασφάλεια. Αυτά που γίνονται λοιπόν σε κοινοτικό επίπεδο Πακής Ένωσης και ακριβώς σε εμά για την άμυνα μέσω της κατάλληλης τεχνολογία. Ρύθμιση λοιπόν, τεχνολογικές πτυχές οι κατάλληλες για να μπορέσουν να ισχύουν αυτά στον εταιρείο χώρο, να εφαρμοστούν και ακόμα κάτι το πρωταρχικό όταν θέλουμε να εργαστούμε για μια πιστοποίηση. Και εκεί όταν υπάρχει περισσότερη δυνατή ανάγκη, μίλησαν και οι ηγέτες κρατών κυβερνήσεων ότι έχει πολύ σημασία αυτό και σε μια συζήτηση μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα δούμε τα εργαλεία που θα έρθουν να μπορέσουν να πιστοποιηθούν όσο γίνεται καλύτερο για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εθνικό επίπεδο. Αποτελούν αυτά τα πράγματα πολύ καλό παράδειγμα πώς μπορούν να συγκλίνουν τη διάφορες μέθοδοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συστήματά της και μετά να δούμε και για πολιτικές αποστολές. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για την μελλοντική χρήση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη που εξοπλίζονται με αυτά ε, και θα ήθελα να ασχοληθώ με τα δύο επόμενα που είναι οι δορυφόροι ε, επικοινωνίας και η κυβερνοασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Νομίζω ότι έχουν να κάνουν με την διαλογική για τους δορυφόρους επικοινωνιών. Έχουμε κάτι που απαιτείται, απαιτείται, είναι απαραίτητο για κάθε μέθοδο επικοινωνίας και ακόμα για κάτι το οποίο χρειαζόμαστε από τώρα το σκεφτόμαστε και για την επόμενη γενιά γιατί εργαζόμαστε μεταξύ των διαφόρων κρατών μέλων Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε αυτές τις δυνατότητες όμως, γιατί διαφορετικά θα γίνουν απαρχαιωμένα τα συστήματά μας. Θα λοιπόν ασχίσουν για τα επόμενα γενιές, να τα λάβουμε υπόψη μας αυτό και για κυβερνητικές ε, χρήσεις. Ε, να είναι κάτι, τα ένα κάτι το ασφαλές σαν σύστημα και να μπορέσει να υπάρχει και μια σύγκληση Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις πολιτικές χρήσεις ε, αλλά και στρατιωτικής φύσεως όπως επίσης και μια τεχνολογική εξέλιξη όπως επίσης και μια βιομηχανική προσπάθεια που απαιτεί αυτή η επόμενη γενιά και ακόμα αυτά στα πλαίσια του κυβερνοασφάλειας και ακόμη για την πιστοποίηση έχουμε μια εντολή του Ευρωπαϊκού από τον Ιούλιο με μια ε, έκθεση έχει ζητήσει, έχουν ζητήσει και θέλουμε για το μέλλον να εργαστούμε για την τυποποίηση, την πιστοποίηση ακριβώς ε, και στο νότο για το Στάνναγκ του ΝΑΤΟ δεν υπήρχε μέχρι τώρα τίποτα. Εντάξει, θα μπορούσε να υπάρξει ένα πολιτικό στάνταρτ πρότυπο και να δούμε την επόμενη διαδικασία την, που θα ακολουθεί για την πιστοποίηση. Ίσως και υβριδικά συστήματα και διαδικά συστήματα μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Και επίσης εκεί που χρειάζονται πρότυπα καθαρά στρατικό από το Στάνναγκ ακριβώς όπως αυτά έχουν καθοριστεί και αυτό σε πλαίσια ας πούμε της Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ασφάλειας ε, και αυτό με την ε, ε, ΑΖΑ σε στενή συνεργασία μαζί της ε, και όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχουν δυνατότητες κοινού προσδιορισμού των αναγκών και μια μη βοήθεια και συνεργασία για την πιστοποίηση. Ακόμα δύο εντολές τρομερά φιλόδοξες και που όπως είπατε κυρία Πρόεδρο μεταξύ της κυρίας Μογκερίνη και του Υπουργού και των Αμήνης συζητήθηκαν πριν από δέκα περίπου μέρες. Πρόκειται για ορισμένες ας το πούμε έτσι παροτρήσεις. Όχι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει. Και αυτή μάλιστα σε ανώτατα επίπεδα ε, από αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων και με τους υπουργούς αμήνους που ένα κώδικο συμπεριφοράς έχουν προσυπογράψει, έτσι. Και συμφώνησαν ε, να, συνεργαστούν σε αυτό ένα policy framework ε, για να στα πλαίσια μιας συνεργασίας, αλλά και πάλι συναντάμε δυσκολίες ε, για το πώς η διοίκηση και αρμόδιες υπηρεσίες θα τα εφαρμόσουν αυτά σε εθνικό επίπεδο, γιατί παραμένουν εθνικού επίπεδου, εθνικής αρμοδιότητας. Και εντάξει, για αυτές τις παροτρήσεις λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο τι λέει. Ε, φορολογικές ας τις πούμε έτσι, non-distorting fiscal measures στα αγγλικά και επίσης άλλα πλαίσια του NSPA. Να υπάρχουν δυνατότητα και για απαλλαγές ε, φορολογικές, ε, αλλά όχι όμως σε προγράμματα τα οποία γίνονται στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού σχεδιασμού και με το Ίδρυμά μας λοιπόν στην εργασία με την Επιτροπή εμείς πετύχαμε μια λύση και νομίζω ότι έχουμε ευθυγραμμιστεί εφαρμόζοντας τους σχετικούς ε, ε, κανονισμούς ας πούμε για το ΦΠΑ και να μπορέσουν να υποφεληθούν και στα πλαίσια του ακριβώς του Ευρωπαϊκού να μπορέσουν να υποφεληθούν και τα προγράμματα με ας πούμε, τριών προγραμμάτων τα οποία προχωράμε. Και στην εντολή επίσης ε, υπάρχει ένας μηχανισμός για μια κοινή αγορά. Κοινή αγορά εξοπλισμού και συζητιέται αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε υπουργού τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να προβλεφθεί. Μην ρευθούμε όμως ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα μια μέρα θα έχει εναρμονιστεί ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο σχεδιασμός αυτός ε, έχει να κάνει και με εθνικό σχεδιασμό και με πολιτικές αποφάσεις, καταλαβαίνετε. Ορισμένα κρατημέλη που εδώ και πάνω από 10 χρόνια εργάζονται για αυτή την εναρμόνιση του σχεδιασμού ε, νομίζω ότι ορισμένοι δεν ακολουθούν ρεαλιστική γραμμή. Άλλοι πάλι έχουν απογοητευτεί από τη εναρμόνιση. Για να δούμε. Πώς θα βρούμε έναν τρόπο. Όχι να εναρμόσουμε το σχεδιασμό της άμυνας παντού. Δεν μου καταφέρνει αυτό να το κάνει το ΝΑΤΟ. Ε, δεν προσπαθεί να το κάνει. Είναι εθνικής αρμοδιότητος. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα από τη στιγμή που θέλουμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα και αυτό κάτω στις καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Έτσι. Αυτό ακριβώς προτείναμε στην συνάντηση των Υπουργών με ορισμένα μέτρα που νομίζουμε ότι τα δέχτηκαν θετικά. Να τονίσω ακόμα κάτι. Το μεγάλο μέρος της οικογένειας της Ευρωπαϊκής ε, δεν θα επανέλθω σε αυτό. Νομίζω ότι συζητήσατε πριν από μένα και το συζητάτε συνεχώς εδώ στην υπεπιτροπή σας αυτό το πλαίσιο το στρατηγικό, τις απειλές, τα μέσα, το τι μπορεί να γίνει. Πώς θα υλοποιηθούν πραγματικά αυτές τις δυνατότητες από τη που είναι πραγματικές, ε, που έχουν να κάνουν με προτοριότητες, τις οποίες συμφωνούν όλοι και άλλα διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και αυτό για να στηρίξουν αυτές τις προτεραιότητες για να μπορέσουμε να υπρασπιθούμε τα συμφέροντά μας και για μια ευμάρεια και λοιπά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παίξουμε και τον κατάλληλο ρόλο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως απαιτείται από την στρατηγική, την πολιτική κοινή ασφάλειας και άμυνας. Να δούμε τώρα στο μέλλον Διότι στο ιδιαίτερα σημαντικού ε, στη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια να κάνω μια εκτίμηση σχετικά με την άμυνα τα μέτρα, τις οδηγίες για την αγορά εξοπλισμού. Η ανάλυση θα πρέπει να είναι λεπτή και βαθιά πάνω σε αυτά τα θέματα και να δούμε από του χρόνου. Και η Επιτροπή Κανονικό το 2016 θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση για να δούμε όλα αυτά μπορούν να προχωρήσουν με με τους στόχους οδηγίας αυτής. Και κάτι ακόμα. Τώρα που έχουμε, είμαστε στα πλαίσια αυτής της πραγματικής πολιτικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η οδηγία να μπορέσει να βοηθήσει μια συνεργασία στην άμυνα, να βοηθήσει και μια ενιαία αγορά, αυτός είναι και ο στόχος. Αλλά μπορεί να συμβαδίζει σε στενή συνεργασία σε θέματα άμυνας, ένας αμοιβαίος χαρακτήρας να το σήμερα όλοι αυτό επιδιώκουμε. Και ακόμα κάτι πολύ σημαντικό για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έρευνα και τεχνολογία. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό εδώ στην Επιτροπή έχετε ιδιαίτερα εργαστεί. Και είστε συνεχώς σε επαφή με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι. Για να δούμε πώς επειδή τα μέσα γίνονται ε, όλα ένα και πιο δύσκολα για λιγότερα προγράμματα. Πώς θα προετοιμάσουμε το μέλλον χωρίς να υπονομεύσουμε ή να θέσουμε να αμφιβόλο την τεχνολογική δυνατότητα στην Ευρώπη γιατί οι βιομηχανίες άμυνας ε, δεν έχουν αγορά ντόπια, άρα λοιπόν ε, απευθύνονται εκτός ευρωπαϊκού χώρου με ορισμένους περιορισμούς αλλά και βάση μεταφοράς τεχνολογίας και αυτές όμως ε, οι μεταφορές τεχνολογίας ευνοούν τους αντιπάλους μας, τους ανταγωνιστές μας. Ε, όχι δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με άλλους, αλλά ε, να μην έχουμε αυτές εμείς τις δαπάνες και με τις χώρες BRICS και με τις ΗΠΑ. Με τις χώρες BRICS ακριβώς έχουμε τεράστιο χάσμα που δημιουργείται τα διάφορα μέσα που έχουμε αναπτύξει στο Ευρωπαϊκό Ιδρύμα Ασφάλεια, Ακριβώ μάμυνα ε, για την έρευνα, την τεχνολογία, τι προσπάθειε οι οποίε καταβάλλονται. Νομίζω ότι χρειάζεται πολλά τα πράγματα να γίνονται συνεργασία με τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, έρευνα, τεχνολογία και η Επιτροπή ήταν πρωτοπόρα σε αυτά, σε αυτό το διοδικό χαρακτήρα βασιζόμενη ε, αεροναυπηγική, στην κυβερνοπροστασία και ε, την ε, προστασία για βακτηριολογικούς, χημικούς πολέμους κλπ. Και επίσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πώς θα έχουμε μια έρευνα για την πολιτική κοινή άμυνας και ασφάλειας. Επίσης η Επιτροπή, η Επιτροπή ανέλαβε μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική σας συγχαίρομαι γι' αυτό για χρηματοδότηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων 2015-2016. Και έτσι να δούμε τις προπασκευές αυτής της τι μπορεί να γίνεται. Πρώτα απ' όλα να μπορούν να δίνονται κονδύλια και να υπάρχει μια συγχρηματοδότηση ανάμεσα στον κοινοτικό προπολογισμό, την δηλαδή και τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη και όλοι οι οργανισμοί εδώ θα πρέπει να συνεργάζονται, να ξέρουν ποιες είναι οι προτεραιότητες. Χρειάζεται και μια συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα προγράμματα έρευνας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εθνικά. Και εμείς θα βοηθήσουμε και ακριβώς νομίζω ότι πραγματοποιήθηκε η πραγματική ανταλλαγή απόψεων και με ένα εργαστήριο μαζί με την Επιτροπή, μια πολύ καλή συζήτηση κλπ που έλαβε χώρα για τους διευθυντή των εξοπλισμών. Για την ε, βιομηχανία τώρα πολύ σύντομα, γιατί πρόκειται για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι ζητάει η βιομηχανία, ζητάει καταρχάς προγράμματα, όχι επιδοτήσεις, προγράμματα. Εναρμόνιση των αναγκών. Ένας πρόσωπο του κλάδου έλεγε χθε στο Βερολίνο ότι χρειάζεται να είναι ενιαίες οι προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και τα προϊόντα. Η εναρμόνιση λοιπόν ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας και εδώ η συνεργασία με την ΕΚΑΦ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Και επίσης αυτό ωφελεί κάθε τύπο βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρομεσαίες το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Άμυνας υφίσταται για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να συγκλίνουμε και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάποιων σχετικών ε, βιομηχανικών παραγωγών των κρατών μελών, κυρίως Κεντρική και ανατολική Ευρώπη που προέρχονται από διαφορετικά συστήματα, πολύ διαφορετικά συστήματα, αλλά που μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του δόγματο ε, τη τεχνολογική και βιομηχανική ικανότητα παραγωγή μας για το μέλλον. Και έχουμε ω εκ τούτου εμεί ειδική δουλειά ξεκινήσει και αναπτύξει για, ε, το δυναμικό βιομηχανική παραγωγή των κρατών τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Κατα, εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί κανεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτή εκφράζεται σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου των Υπουργών έχει επιβεβαιωθεί από, τους, από την νέα ηγεσία των θεσμικών οργάνων, την κυρία Μογκερίνη, τον κύριο Γιουνκέρ. Προτεραιότητα λοιπόν θα δοθεί στην άμυνα. Ο κύριος Τούσκ αναλαμβάνει την προπαρασκευή του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλέον λοιπόν το ζήτημα δεν είναι η συμπληρωματικότητα των προσπαθειών με τον ΝΑΤΟ, γιατί αυτή είναι απόλυτη, επιβεβαιώνεται στην Σύνοδο της Ουαλίας στη Σύνοδο των Μελών του ΝΑΤΟ θα επιβεβαιωθεί από το Προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι εταίροι και οι παράγοντες να συνεργάζονται και εγώ μια και κάπου στα μέσα Ιανουαρίου θα ε, έχω πια αποχωρήσει. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστώ θερμό ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως τα μέλη της Επιτροπής σας για την εξαίρετη συνεργασία και που πιστεύω και, να εκφράσω, και θέλω να εκφράσω την ευχή επίσης να μετατραπεί αυτή η συνεργασία ε, σε μια ακόμη πιο ε, εντατική συνεργασία με τον διάδοχό μου, γιατί θα πρέπει όχι μόνο να γίνει η προεπαρασκευή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και τις συνέχεια μετά από αυτό, όπου ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ε, είναι πολύ πιο σαφής ως προς τις δημοσιονομικές αλλά και κανονιστικές ρυθμίσεις και επαφάσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αρνό. Ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. και μπορούμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων με τον κύριο Νάρτ πρώτα που δεν μπόρεσε νωρίτερα να λάβει το λόγο. Δεν έχω ερώτηση λέει ο κύριος Νάρτ. Η κυρία Λούζιν. Μπορώ να αρχίσω τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις που γέννησε αυτή η παρουσίαση. αφόρμητες ερωτήσεις και μια-δυο ερωτήσεις για διευκρίνηση περισσότερο. Καταρχάς λοιπόν, μια και μιλάτε για πολιτική βούληση. Ξέρουμε ότι πολλής λόγος γίνεται για το γεγονό οτι ότι πολλοί άριθμα κράτη-μέλη θέλουν ενίσχυση, ε, μάλλον είναι επιφυλακτικά έναντι της ενίσχυσης της ΔΕΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αμήνας. Μπορείτε να μα πείτε ποια είναι αυτά τα επιφυλακτικά κράτη-μέλη και τι αναλογίες έχουμε σε αυτή την ε, ισορροπία δυνάμεων. Από πλευρά τη Γερμανία υπάρχουν πολύ ισχυρά μηνύματα προ την κατεύθυνση αυτή. Και θα ήθελα να αναφέρω κάτι που διάβασα σε ένα εσωτερικό έγγραφο του Bundestag της Γερμανικής Βουλής όπου λέγεται ότι με την υποστήριξη των κρατών μελών θα πρέπει η υπηρεσία στο μέλλον να είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και για μεγάλα προγράμματα προμηθειών ε, και για ε, θέματα εξοπλισμού με τη μορφή παραδείγματι κινήτρων φορολογικών, απαλλαγή από τον φόρο προσθέμενης αξίας σε περίπτωση προμηθειών ε, ή ανάληψη κάποιων δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή μας έχουν, δεν ξέρω αν είσαστε και εσείς ενημεροί, Έχουμε συζητήσει και με έντονη αντιπαράθεση σε σχέση με την ε, απαγόρευση χρηματοδότησης μέσων με στρατιωτική χρήση, προϊόντων στρατιωτικής χρήση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτή την απόφαση. Επίσης, όταν μιλάτε για μεγαλύτερο ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας για τις ε, προμήθειες και όταν γίνεται λόγος για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτών των δραστηριοτήτων πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτό στην πράξη και πώς μπορεί να συνάδει με την απαγόρευση παραδείγματι της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων Όταν ας πούμε έχουμε τα προϊόντα διπλής, διαδικής χρήσης, διπλής χρήσης στρατιωτικής και μη στρατιωτικής, στα οποία αναφερθήκατε εσείς και που μπορούν να αποτελέσουν όπως λέτε μία ε, ευκαιρία για λύση της, ε, των προβλημάτων. Αυτή η απαγόρευση που προκύπτει από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθεί υπόψη ή καθόλου. Έχει σημασία η έρευνα είναι σαφές από την συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση έρευνας για στρατιωτικό σκοπό από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό. Και τι ρόλο μπορείτε να διαδραματίσετε εσείς ως υπηρεσία ε, στη, στα μεγάλα αυτά έργα και τις προμήθειες. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο στους συναδέλφους να ξανασκεφτούν καλά ποιες είναι οι επόμενες τους ερωτήσεις και θα παρακαλέσω τόσο την κυρία Αρνούσο και τον στρατηγό Παλομερός να δώσουν απαντήσεις σχετικές ε, με, τον, με τις δυνατότητες για την καταπολέμηση του κύβερνο πολέμου. Δύο υπηρεσίες. Μία εδρεύει στο Ταλίνο, άλιστα έχει συσταθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μετά τη μεγάλη εκείνη κυβερνοεπίθεση βάρος Εστονίας το 2007 εάν δεν με απατάει μνήμη μου. Και υπάρχει και ένα κυβερνοκέντρο στη Χάγη. Πώς αξιολογείτε τις δυνατότητες των δύο αυτών κέντρων για την αντιμετώπιση του κυβερνού πολέμου. Και επίσης, κυρία Αρνού, τι θέλετε να πείτε για τον τομέα αμήνης των νέων κρατών μελών. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες ιδέες, όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων είμαι βεβαία ότι πολλές είναι και καινοτόμες και ανταγωνιστικές. Μάλιστα υπάρχουν και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και μεγαλύτερες. που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας. Αλλά υπάρχουν και άλλες που είναι πολύ παραδοσιακών δομών. Δεν είναι ακόμη δηλαδή ενιαία εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος. Τι ευκαιρίες βλέπετε για αυτές τις επιχειρήσεις για ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Ράντος. Κύριε Πρόεδρε, το 2008 μέρος των κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων στην τεχνολογία. Το ποσοστό μάλλον αυτό ήταν 16% οι μελητής. Ως τη συνολική δαπάνη δηλαδή για έρευνα και τεχνολογία. Την εποχή εκείνη, η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είχε θέσει στόχο το 20% του συνόλου δηλαδή των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία. Δεν ήταν και πολύ φιλόδοξος ο στόχος και θεωρώ ότι κυρία, για την κυρία Αρνό στο τέλος πλέον της θητείας της η ερώτηση είναι ε, απαραίτητη. Ποιο είναι το ποσοστό σήμερα επί του συνόλου δηλαδή των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία. Πάρα Παρακαλώ. Κύριε Γενικέ. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση της κυρίας Λέζινγκ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση και πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στην ε, Γερμανική Βουλή, στην Bundestag. Δεν μπορώ φυσικά να τη σχολιάσω καθώς αποτελεί η εθνική αρμοδιότητα 100%. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω με ειλικρινή διάθεση είναι ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης το λιγότερο τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Πρέπει να καταλάβουμε όμως το γιατί. Εάν δείτε τα κύρια, τα μεγαλύτερα προγράμματα, τις βασικές μας δραστηριότητες. Θα δείτε ότι η Φιλανδία, στην θαλάσσια επιτήρηση, η Αυστρία, στην αποτελεσματική, στο, στο σύστημα προμηθειών, η Ιρλανδία, στην εκπαίδευση, είναι επικεφαλής. Αυτές οι χώρες είναι επικεφαλής σε αυτά τα προγράμματα και ξεχνώ και άλλα προγράμματα βεβαίω που δεν είναι το παρόντος. Και η Ολλανδία βεβαίω είναι μπροστά σε πολλά προγράμματα. Ένα αέριο ανεφοδιασμός, ανεφοδιασμός σε πτήση, Συμμαχικέ δυνάμεις στο Αφγανιστάν, συστήματα αναγνώριση κλπ. Για μένα, μετά από τέσσερα χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό απο μικρομεσές μικρομεσαίες, από μικρομεσαία κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμυνάς. Ήδη τρεις βαλτικές χώρες, αλλά και άλλες χώρες ακολουθούν στον ίδιο δρόμο. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινεί Ακόμη δεν έχει αγκαλιαστεί η υπόθεση από τα μεγαλύτερα κρατημέλη. Γι' αυτό και είπα, χρειαζόμαστε κίνητρα. Τώρα κάποια πράγματα ο καθένας μπορεί να τα κάνει μόνος του η συνεργασία στον τομέα της άμυνας ε, δεν είναι, σίγουρα δεν είναι φυσική, δεν προκύπτει αυθόρμητα θα έλεγα. Τα Υπουργεία Μήνης δεν έχουν φτιάξει για αυτή την υπόθεση. Ε, και οι συνήθεις ερίδερες είναι αν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, θα το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό βλέπω τέσσερα χρόνια τώρα. Λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι κατά περίπτωση και κατά βούληση. Είναι ένας μηχανισμός τον οποίο επιφορείται κάποιοι εάν και εφόσον. Εάν και εφόσον. Εάν δηλαδή τα ωφέλη είναι άμεσα και ορατά. Αν μπορούν δηλαδή να αξιοποιήσουν και να αποφελθούν κάτι μέλη από την τεχνική ή άλλη τεχνογνωσία κάποιου άλλου. το λέω και όχι επειδή είμαι στο τέλος της εντολής μου, ο οργανισμός αυτό αξίζει τα περισσότερα προγράμματα στην έρευνα και την τεχνολογία, πρέπει να σας πω, είναι με τη συμμετοχή τριών-τεσσάρων χωρών το πολύ. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Είναι κρίμα από την άλλη πλευρά που ακόμη και σήμερα τα μεγάλα κρατημέλη δεν δείχνουν το δρόμο. Πρωτοπόρα είναι τα μικρά κρατημέλη. Και εδώ χρειαζόμαστε επενδύσεις στους πιο κρίσιμους τομείς. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και στα μεγάλα κρατημέλη να συμμετάσχουν όπως και στην βιομηχανική και αμυντική υποδομή. Υπάρχουν τομείς, ε, δορυφόροι, ενέριος, ε, ανεφοδιασμό, ανεφοδισμός, σε κλπ. Εκεί υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει και εκεί πρέπει να δείξουμε ακριβώς την αλληλεγγύη μας με τα μικρότερα κρατημέλη και να συνταχθούμε στην κοινή προσπάθεια. Ευελπιστώ ότι ότι ο διαδοχός μου θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει όλα αυτά όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Νέα Επιτροπή και στην Επιτροπή της Bundestag για την άμυνα. Αυτά. Παρόμοιε συζητήσει είχαμε σε διάφορα άλλα εθνικά κοινοβούλια. Την περσμένη εβδομάδα ήμουν στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Έχω προσκληθεί πολλέ φορέ στη Βουλή των Λόρδων, για να συζητήσουμε το, τη σκοπιμότητα το κατά πόσο να αξίζει να είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας κλπ. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες παρανοήσεις, κάποιες παρεξηγήσεις και γι' αυτό καλό είναι να γίνονται απευθείας συζητήσεις με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές άμυνας στην κάθε χώρα. Έχει γίνει αυτό βέβαια και πρέπει να ξαναγίνει. Όλα τα κρατημέλη και τα μεγάλα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Πολλές φορές μας λένε τα κρατημέλη, μα πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα, είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Όντως, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός και μόνο, που λειτουργεί όντως αλλά Αλλά Κάποιοι πρέπει να δείξουν το δρόμο. Αυτοί που ακόμη δεν έχουν πιστεί, τα μεγάλα κράτη, που είναι λίγο επιφυλακτικοί, πρέπει να μπουν στη θέση του οδηγού και να δείξουν το δρόμο. Να πάρουν πρωτοβουλίε. Τώρα, για την έρευνα. Όλο και περισσότεροι τομεί είναι τη λεγόμενη διτή χρήση. Και εδώ θέλω την υποστήριξη τη επιτροπής σας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπερασματά του και στις διάφορες εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου λέγεται ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αυτό το λένε και οι συνθήκες. Χρειάζεται λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό ακούω παντού και πάντα. αυτός είναι ο σκοπός και πάμε. Ω πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τον κυβερνοχώρο, ο τέτοιος Παλαιμερό θα μα πει για το Ταλίν και το NCIA. Το θέμα πάντως το συζητήσαμε με το Τάλιν, το και το Ταλίν, για να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία τους, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχουμε επίσης πολύ καλή συνεργασία με το NCIA, που είναι αρμόδιο, κατά κύριο λόγο, για την προστασία των δομών του νατός. Τιμός. Θέλουμε απόδοση αποτελεσματικότητα, αλλά είμαστε και ρελιστές όσον αφορά τα του κυβερνοχώρου και θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εκπαίδευση και την ενημέρωση, το NDIA δουλεύει στην ε, Λάρισα και επίση έχουμε πρωτοβουλίε στην έρευνα και την ανάπτυξη όπου τα κράτη-μέλη ε, έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν από κοινού. Κάναμε τα πρώτα βήματα και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα κάνουμε και τα πρώτα πραγματικά ουσιαστικά βήματα. Και εδώ και πάλι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, πολλή διστακτικότητα και στον τομέα του κυβερνοχώρου, αλλά και εδώ πρέπει να προχωρήσουμε. Επίσης, σταδιακά βεβαίως, φτιάχνουμε και kit τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν επί τόπου οι αποστολές μας. Τώρα για την βιομηχανία του EDA να δουλεύει για τη βιομηχανία, την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το ξαναλέω. Και όχι μόνο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει αλλά και για τις μεγάλες βιομηχανίε. Λαμβάνοντας υπόψη τι δημορφίε και των νέων κρατών μελών. Διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν ωφελή για όλου τώρα που όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να υλοποιήσουν το νέο πακέτο χωρίς αναγκαστικά σε όλες τις περιπτώσεις ε, αντισταθμιστικά ωφελήματα. Τώρα, ως προς το άλλο ερώτημα, κύριε Δεν μπορώ να απαντήσω αποστήθουσαν και έχετε δίκιο, ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να εξηγήσω, να περιγράψω την κατάσταση. Παντώ ναι, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Αν και δεν ευθύνουμε εγώ, αλλά ανησυχούμε για τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. Σίγουρα δεν έχουμε πετύχει το 20% και είμαστε σε κάθε περίπτωση μακριά από εκεί που ήμασταν το 2008. Πρέπει πάση θυσία να βρούμε μία λύση προκειμένου. Γιατί? Διότι ήταν περικόπτη σε έναν αμυντικό προπολισμό αυτό που κάνουν όλα τα κρατημέλη, ακόμα και αν αυτό αφορά προσωπικό, πηγαίνουμε πίσω. Οι οικονομίες δεν γίνονται αισθητέ αμέσως, γι' αυτό το πιο εύκολο για να έχει άμεση οικονομία είναι να περικόψει προγράμματα έρευνα και εξέλιξη. Και η επίπτωση στη βιομηχανία είναι άμεση δυστυχώ. Είναι διπλό το πλήγμα. Με τη σειρά τη δεν επενδύει στην έρευνα ούτε η βιομηχανία. Οπότε πρέπει να κάνουμε το αντίθετο, να δώσουμε κίνητρα για επενδύσει, στην έρευνα και την ανάπτυξη. Θα ξαναπώ φορολογικά μέτρα, φορολογικά κίνητρα, αυτά χρειαζόμαστε. Κίνητρα στην περίπτωση συνεργατικών σχεδίων. Αυτό είναι ο δρόμος που προσπαθούμε να ανοίξουμε και με τη συμμετοχή ευελπιστώ του ιδιωτικού τομέα. Αυτό προσπαθεί να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του σχεδίου επενδύσεων. Ναι, για να προσθέσω και για το κυβερνό πόλεμο, είναι προφανώς μια από τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, θα το αντιλαμβάνονται οι πάντες ασφαλώς και χρειαζόμαστε κάθε δεξιότητα, ικανότητα, γνώσεις, προσπάθειες, μελών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, του ιδιωτικού τομέα, του, της βιομηχανικής παραγωγής, των λοιπόν επιχειρήσεων για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες αυτές προκλήσεις και τον κίνδυνο αυτό που επιτρέπει, όχι μόνο όσον αφορά την άμυνα, αλλά και την κοινωνία γενικότερα και την παραγωγή και πολλούς άλλους τομείς. Τι κάνουμε λοιπόν όσον αφορά το ΝΑΤΟ. Στόχος μας είναι να προστατέψουμε το σύστημα διοίκησης και ελέγχου να είναι ασφαλές, γερό και αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο η υπερασία ε, πληροφοριών της Χάγης του ΝΑΤΟ ε, εργάζεται και η δουλειά μας είναι τέτοια που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραματίσει το ρόλο της. Το έχω ήδη αναφέρει και εκθέσει αυτό. Ο κυβερνοπόλεμος όμως είναι και πανταχού παρόν πρέπει να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε μια κυβερνοαπειλή σε έναν τομέα και τη λησμονούμε στις λοιπές εξελίξεις γιατί βρίσκεται σε κάθε εξέλιξη, κάθε είδους εξοπλισμού. Εάν πάμε να δούμε παραδείγματι τις μεγάλες αεροπορικέ ε, αεροπορικές το κυβερνό το έχουν στο επίπεδο των ενδιαφέροντός τους. Τα δε κέντρα ε, υπεροχής αναπτύσσονται στα κράτη-μέλη με μια συνεννόηση, με μια συναντήληψη, χωρίς να ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αναπτύσσονται σαν κέντρα υπεροχής για να παρέχουν υπηρεσίες, κατάρτιση, έρευνα, τεχνολογία, δεξιότητες, οτιδήποτε είναι η ειδικότητα τους, ο τομέας δραστηριοποίησης τους, σε επίπεδο ε, ΝΑΤΟ. Το ειδικά δε το κέντρο αυτό που βρίσκεται στην Εστονία για το κυβερνό έγκλημα έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Ήταν πολύ περήφανο για αυτό το κέντρο και προσπαθούμε να αντλήσουμε στο δυνατόν περισσότερα ωφέλη από αυτή την επένδυση, να ανοιχτό στους εταίρους και γιατί να μην μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Έχουμε οργανώσει, όπως είπα και νωρίτερα πρόσφατα, μια μεγάλη επιχείρηση του ΝΑΤΟ με 900 συμμετέχοντες από 18 διαφορετικές χώρες, κυβερνοσυμμαχία, ε, υπεύθυνους για κυβερνοάμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης παρόντες. Μια μεγάλη άσκηση. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ε, γνώση μας, την ευαισθητοποίησή μα και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο το να γίνονται και τέτοιου είδου ασκήσει. Μέχρι τώρα επικάλυψη δεν έχω δει. Μάλλον ελλείψει διαπιστώνω. Παρά επικαλύψει. Η πρόεδρο ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώνεται νομίζω έτσι το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης και για άλλη μια φορά Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κλωτ Φανσαγνό και τον στρατηγό Ζων Πολ Παλομερός που ήρθαν στη συνεδρίαση μας. Θα σας παρακαλέσω, αγαπητοί συνάδελφοι, να μείνετε εδώ. Θα διακόψω μόνο για δύο λεπτά για να χαιρετήσω, να ξεπροβοδήσω ε, τους προσκεκλημένους μας και θα πάρουμε μετά στα λοιπά θέματα. Την ενημέρωση δηλαδή για την πρόσφατη κοινοβουλευτική συνέλευση της κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και παρουσίαση από τον κύριο Ποπόφσκι αναπληρώτη Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τα θέματα του Υπουργείου των Εξωτερικών. Ευχαριστώ. started explaining to the others what you did in Oh, shit. Ladies and gentlemen, please be seated once more. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε και πάλι. Το επόμενο θέμα. στην ημερήσια διάταξη είναι ενημέρωση για τις δραστηριότητες της πρόσφατης κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Καλωσορίζω την κυρία Εύα Καηλή, επικεφαλής πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με το ΝΑΤΟ και την παρακαλώ να μας κάνει την παρουσίαση, να μας δώσει τις πληροφορίες της για τις εργασίες της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Στη Χάγη το Νοέμβριο από τις 21 στις 24 του μηνός. Thank you very much, uh, Ms. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η, Ευρωπαϊκή, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σχέση με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, όπως είπατε κι εσείς, ναι, και ήσασταν και παρούσα μάλιστα έλαβε μέρος στην 60η ετήσια κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ από τις 21-24 Νοεμβρίου στην ΧΑΚ. Είχα την ευκαιρία λοιπόν μαζί με εσάς να συμμετάσχω στις δραστηριότητες όλων των συνεδριάσεων επιτροπών και στην Ολομέλεια. Λάβατε φαντάζομαι όλη την έκθεση που εκδώσαμε κατόπιν τη συνεδριάσεω αυτή. Είχαμε πολλέ ευκαιρίε να παρακολουθήσουμε συζητήσει για διάφορα θέματα σχετικά με τι φυστάμενε απειλέ και προκλήσει για την ασφάλεια όχι μόνο τη Ευρώπη αλλά και πέραν αυτή συζητήσεις οι οποίες επικεντρώθηκαν στις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, ιδίως τις, τα, τα μέτρα επιβεβαίωσης καθησυχασμού και υποστήριξη εταίρων, εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, κατάσταση στην Ουκρανία που απασχόλησε το περισσότερο διάστημα νομίζω, σχέση με τη Ρωσία, ασφάλεια και πολλά άλλα. Οι συστήσεις και εκθέσεις ε, Στράφηκαν επίσης γύρω από θέματα ασφάλειας ε, και εξωτερικά σύνορα και ενέργειας ε, στα εξωτερικά σύνορα, θέματα που μας απασχολούν και εμάς τακτικά. Είδαμε παρουσιάσει από τον ε, Ολλανδό μεταξύ άλλων Υπουργό και από διάφορα Ινστιτούτο, Ολομέλη, ο κύριος Στόλτερμπερκ έκανε μια ομιλία στην οποία υπογράμμισε πολλά ζητήματα ασφάλειας, απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις. Εγώ παρακολούθησα ιδιαίτερους εργασίες πολιτικής Επιτροπής της Επιτροπής ε, επίσης Επιστήμων και Τεχνολογίας. Ξέρω ότι και εσείς ολόκληρη ημέρα παρακολουθούσατε όλες τις επιτροπές. Το πιο σημαντικό νομίζω ήταν το θέμα της ασφάλειας, ε, της δυναμικής ασφάλειας στα νοτιοτολικά σύνορα της Ευρώπης, προοπτικές διατλαντικής συνεργασία, ασφάλεια ενεργειακή, ε, ενεργειακή αγωγή για την Ευρώπη και είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα ασφάλεια, ζητήματα κοινού, κοινά. Η επόμενη ευκαιρία νομίζω θα έχει, την επόμενη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε όλοι και οι δέκα της αντιπροσωπείας και αν έχω λίγο ακόμα χρόνο, σας ευχαριστώ θερμά, θα ήθελα να εστιαστώ σε ένα-δύο ζητήματα με κάλου ενδιαφέροντος. Η εταιρική σχέση του ΝΑΤΟ και η πολιτική ανοιχτών θυρών, η ασφάλεια ενέργειας στην Ευρώπη και οι οικονομικές κυρώσεις, οι συνέπειες των οικονομικών κυρώσεων της Ρωσίας προς τη Ρωσία, μια και είμαστε οι εγκύτεροι προς τα εδάφια αυτά γείτονες, κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν, τεχνολογία, πυρηνική ενέργεια, ασφάλεια. Αυτό που ο κύριος Στόλτπερκ τώρα. Βλέπουμε ότι θεωρεί πως κύρια προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί ο προπολογισμό και υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσει που είναι απαραίτητε για να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίε. Αντιλαμβανόμεθα ότι η Ρωσία ήταν πιο καλά προετοιμασμένη, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε κατά το 2% του ΕΠ, ε, το, έως το 2% του ΕΠ το ποσοστό για τον ΝΑΤΟ. Επίσης εξελέγει νέος ε, πρόεδρος ε, από το Κογκρέσο για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Υποστήριξαν οι πάντες τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της Συνόδου της Ουαλίας. Ανησυχία εκφράστηκε για την για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι σαφές ακόμη μέχρι πού μπορεί να επεκταθεί, κανείς δεν είναι αρκετά προετοιμασμένος. Ενδιαφέρον θέμα και το οποίο δεν περιμέναμε να ακούσουμε στο ΝΑΤΟ, πιστεύω. Ήταν η έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για καλύτερη επεξήγηση και ανάλυση των επιχειρημάτων της TTIP που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ένωση και θα συνεχίσω ακόμη για ένα-δύο δευτερόλεπτα εάν έχω την υπομονή σας. Συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμαχία μας. Υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση λιθών. Λοιπόν, καλύτερη ε, καλύτερο επιμερισμό των βαρών και των ευθυνών. Δεν υπάρχουν πια σύνορα, όλοι πρέπει να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο η Πολωνία έχει φτάσει στο 2%, όπως άλλωστε και το Ηνωμένο και η Ελλάδα. Και μια ακόμη χώρα έχει φτάσει στο 2% επί του ΑΕΠ. Οι υπόλοιπε χώρες όμως πρέπει να κάνουν περισσότερη προσπάθεια. Ενδιαφέρον επίσης ήταν ότι εκφράστηκε συμφωνία για τη συνεργασία στην ε, πυραυλική άμυνα με ε, αγορές συστημάτων. Νομίζω αυτά. Ήταν ο Στόλτερμπερκ πιο συγκεκριμένα είπε ε, και σαν παράδειγμα όμως είναι σημαντικό ότι το ΝΑΤΟ έχει πιο πολλές έχει πενταπλάσεις ενέργειες αποστολές τώρα από ό,τι στο τέλος στις αρχές του, προηγούμενου, του φετινού χρόνου αποστέλει ε, πολεμικά πλοία στη Βαλτική γενικά θα αυξήσει πολύ γρήγορα την ανά, τις αναπτύξεις ε, Υπάρχουν ζητήματα ανθρωπιστικών κρίσεων, Ουκρανίας, υποστήριξη στο Αφγανιστάν, που εξέφρασε και συνοδός της Ουαλίας, ε, απειραυλικής άμυνας, με βαριστικούς πυράβλους. Ήταν ενδιαφέρουσα λοιπόν η συνεδρίαση και νομίζω ότι και για το μέλλον μπορούμε να ε, δούμε ε, πώς μπορούμε να εκφράσουμε την, ορα, την, την τοποθέτησή μας, τη βούλησή μας, να είμαστε και πιο ορατοί σε αυτές τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις και φυσικά αυτό υπό τη δική σας καθοδήγηση και βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα σύνοδος. Ακούσαμε όχι μόνο υψηλά εστάμενους πρόσωπος του ΝΑΤΟ αλλά και αξιωματούχους της Ολλανδικής Κυβέρνησης και εμπειρογνώμονες με γνώση πολύ σημαντικών θεμάτων. Ακούσαμε για τον ρόλο του Ισλαμικού κράτους, για τις ε, εσωτερικές απειλές για την ασφάλεια των κρατών μελών. Πολύ ενδιαφέρουσε επαναλαμβάνω παρουσιάσεις, χάρη στι οποίε σήμερα με μια γενικότερη εικόνα. Ακούσαμε επίση ενημέρωση για τη σύμπραξη την ειρήνη. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Οπότε, ε, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πιστεύω ότι χάρη σε όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει την παρουσία του και πιο στις κοινοβουλευτικές συνόδους του ΝΑΤΟ. παρόμοια εμπειρία έχουν πολλοί συνάδελφοι εδώ, στις τη κυρία Μογκερίνη. Αυτό ήταν το μέα τη το Εθνικό Κοινοβούλιο, όπως και ο δικός μου άλλωστε. Θεωρώ ότι αυτές οι συνδίκε και οι έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο κύριος Κίρτσος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλύψατε το θέμα και οι δύο πιστεύω. Απλώς να προσθέσω ότι όλοι ήμασταν ενωμένοι αναγνωρίσαμε την ανάγκη να περιορίσουμε τη μείωση της συρρήκνωσης των αμυντικών προπολογισμών. Βεβαίως δεν άκουσα και πολλές δεσμεύσεις αύξησης των αμυντικών προπολογισμών. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να μειώνουμε τους προπολογισμού μας για την άμυνα. Όλοι ήταν υπέρ της ενίσχυσης της διατλαντικής σχέσης, που σημαίνει ότι εμείς οι Ευρωπαίοι κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε στον επιμερισμό των βαρών, γιατί οι Αμερικανοί δαπανούν πολλά, που νομίζω τρία τέταρτα του συνόλου του αμυντικού τους προϋπολογισμού Θέλουμε επίση να βελτιώσουμε την ποιότητα των ενόπλων δυνάμεων, να ξοδέψουμε, αλλά να ξοδέψουμε σωστά. Και να κοιτάξουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις Βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία. Ομόφωνη ήταν η διάθεση να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ρωσία για την Ουκρανία Όλοι είπαν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την έλλειψη σταθερότητας στην λεγόμενη γειτονιά μας. Δύο σχόλια αρνητικά, αν μου επιτρέπετε, για να γίνει και πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πιστεύω ότι δεν αναλύσαμε τον ρόλο της Κίνας στη συζήτηση των παγκοσμίων προκλήσεων, γιατί είχαμε άλλες προτεραιότητες. Η Κίνα ίσως μας φαίνεται πολύ μακρινή η άποψή μου είναι όμως ότι κερδίζουν στρατηγικά πλέον εκτίματα, ιδιαίτερα μετά από την κρίση στις σχέσεις με τη Ρωσία. Οι εμπειρογόμενες πάντως ήταν ε, εξαιρετικοί Πρέπει να πω, πολλοί από αυτούς δεν σκέπτονται όπως εμείς ας πούμε στον τομέα των οικονομικών κυρώσεων το κόστος για την δυτική οικονομία αλλά και για την ρωσική οικονομία ή για την ενέργεια. Εκεί ακούσαμε διστάμενες απόψεις και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μας έδειξαν δηλαδή προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Πολύ ωραία. Συζήτηση. Ποιο θέλει το λόγο. Συμφωνώ ότι συζήτησαμε μάλλον αυτά που προανέφερα, όντως. Πιστεύω ότι ότι δεν συζητήθηκε την επόμενη φορά να καταγράψουμε αυτά που ενδεχομένω θέλετε να συζητήσουμε την επόμενη φορά και αυτά που θέλουν και οι άλλοι συνάδελφοι να συζητήσουμε για την επόμενη φορά. Μπορεί να είμαστε περισσότεροι, να είμαστε δέκα. Να προετοιμαστούμε όμως πριν ε, θέσουμε τα θέματα. Μπορούμε να ζητήσουμε να γίνει συζήτηση για την Κίνα και όλα αυτά που είπατε στην ετήσια σύνοδο. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ευχαριστώ και τους δυο σας, και την κυρία Καηλή και τον κύριο Κίρτσο. Α, ο κύριος Νάρτα θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, σύντομα στη συνάντηση έγινε ε, μια ανάλυση αυτής της κατάστασης που δεν μπορεί να είναι διαφορετική για τη διαφορά αυτή Ρωσίας και Ευρώπης για ένα άξονα εντελώς προβληματικό και επικίνδυνο άξονα όπως ακριβώς ένα άξονα ρωσοκινέζικο ε, εξετάστηκε αυτό το ενδεχόμενο Όντως, ακούστηκαν σχόλια για τα σχόλια των εμπειρονομών. Ε, η σύνοδος είναι βεβαίως ε, σύνοδος ε, βουλευτών και αυτόν η γνώμη περισχύει. Αυτές καταχωρούνται στις εκθέσεις και τα ψηφίσματα. Τα κείμενα αντικατοπτρίζουν την κυρίαρχη άποψη μεταξύ βουλευτών των χωρών του ΝΑΤΟ. Να κλείσουμε νομίζω, ήρθε η ώρα. Ευχαριστώ το Προεδρείο της ΔΙΝΑΤ για την συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους. Οπότε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Καλώς ήρθατε κύριο Ποπόφσκι. αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τη ΕΕΔ. Ενημέρωση σχετικά με το Συμβούλιο Εξωτερικών Παθέσεων τη 18η Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η συνάντηση 18 η Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η συνάντηση 18 Νοεμβρίου ήταν μια πρώτη συνεδρίαση των Υπουργών Αμήνη επί, ε, υπό την Προεδρία της Νέας Αντιπροέδρου και είπα τη εκπροσώπους εξωτερική πολιτική. Ήταν μια πρώτη ευκαιρία για να επιβεβαιώσει αυτό που είχε πει και εδώ στην ακρόαση η κυρία Μογκερίνη το ενδιαφέρον τη για τα θέματα τη άμυνα και τη ασφάλεια και τη βούλησή τη να διαδραματίσει ρόλο και ω ε, είπα εκπρόσωπος αλλά και ω επικεφαλή τη ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνη και ασφάλεια και βέβαια να δραματίσει το ρόλο τη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεδρίαση ω ήθιστε ξεκίνησε με την ε, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας και την παρουσίαση των συμπερασμάτων της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου του 2013. Η υπηρεσία παρουσίασε κάποιες λεπτομέρειες σχέση με, δημοσιονομικούς και οικονομικ... δημοσιονομικά και οικονομικά κίνητρα στο χώρο της άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα ζήτημα που είναι εν είναι αυτό της εξαίρεσης ε, τις απαλλαγές από το ΦΠΑ για κάποια προγράμματα στο Βέλγιο, μπορεί όμως να ακολουθήσουν και άλλοι. Και υπήρξε κάποια συζήτηση για τα προγράμματα ε, αποτροπής που σας είναι γνωστά και άλλες ζητήματα που συζητήσατε σήμερα με, τον, ε, με την ε, Γενική Διευθυντρία της Υπηρεσίας σήμερα. Επίσης, Έγινε μια παρουσίαση από τον νέο Επίτροπο, τον υπεύθυνο για θέματα βιομηχανίας, ε, την νέα Επίτροπο Μπινκόφσκα για θέματα βιομηχανίας που έχει στο χαρτοφυλάκιό της και την αμυντική βιομηχανία. Άρα περιέγραψε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την έρευνα διαδικής χρήσης, στρατιωτικής και μη στρατιωτικής δηλαδή, καθώς και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που είναι μια συγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης για έρευνα σχετική με την ΚΕΠΑ. Αυτό ανακοινώθηκε, είχε ανακοινωθεί μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη του Συμβουλίου ε, και είναι μια συνεχιζόμενη δουλειά, είναι μια γραμμή δράσης θα λέγαμε. Η συνεδρίαση λοιπόν η ίδια του Συμβουλίου με παρουσία όλων των κρατών μελών ακολούθησε και ήταν μια πάλι μια πρώτη φορά όπου είδαμε προσκεκλημένο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος έτυχε πολύ καλή υποδοχή, τον χειροκρότησαν και όλο στο τέλο της συνεδριάσεως. Η ατμόσφαιρα δηλαδή στι συζητήσεις ήταν ε, πολύ καλή, πρέπει να πω. Πριν από την άφηξή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ χρειάστηκε η Γραμματεία να ασχοληθεί με το ακανθόδε ζήτημα και κάθε χρόνο Μα προκύπτει το ίδιο ε, θέμα συζήτηση, δηλαδή του προπολογισμού της ε, υπηρεσίας αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πατή εκπρόσωπη, για άλλη μια φορά εμφανίστηκε βέβαια η διαφωνία. Ε, η υπατή εκπρόσωπος πρότεινε μηδενική αύξηση, θα ήταν η πέμπτη φορά, πέμπτος χρόνο σε σειρά. Δεν έγινε δεκτή η πρότασή της, με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχιζόμενη μείωση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής πάγικες Υπηρεσίας ε, Αμήνης. Πάντως ε, είπε η εκπρόσωπος ότι πρόκειται τη συζήτηση αυτή να την αναπτύξει ε, πιο ουσιαστικά στην, για την επόμενη χρονιά. Επίσης η Στρατηγική Επιτροπή με τον Πρόεδρό της τοποθετήθηκε για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις ξεκινώντας μάλιστα με την απόδοση τιμών και μνημόνευση ενός στρατιώτη Γάλλου που έχασε τη ζωή του λόγω ελονοσίας. Συζήτηση έγινε για το Μαλί, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αταλάντη. και την αποστολή της Βοσνίας, στη Βοσνία Ζεβοβίνη. Η υπάτη εκπρόσωπος επιβεβαιώνει ότι σκοπεύει να ε, επισκέπτεται στον δυνατόν τις αποστολές ε, και επιχειρήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλωστε έχει ξεκινήσει ήδη, έχει πάει στη Γιούπολ Κόξ της Ραμάλα όταν επισκέφθηκε τις προάλλες ε, τη Μέση Ανατολή. Θα ακολουθήσει μια επίσκεψη την Παρασκευή αυτή στη Βοσνία όπου ελπίζουμε πως θα έχει και την ευκαιρία να συνομιλήσει με στρατιώτες Ευρωπαίους εκεί. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, αλλά ξέρουμε ότι αυτή είναι η πρόθεσή της. Τελευταία στιγμή έγινε και μία προσθήκη στα συμπέρασματα του Συμβουλίου, όσο θα την έχετε δει. Ένα αίτημα προς την επατή εκπρόσωπο να παρουσιάσει μια αντίληψη, μια ιδέα διαχείρισης κρίσεων σε σχέση με την κεντροαφρικανική ε, ε, δημοκρατία. Η U4CAR έχει δει την επέκταση των δραστηριοτήτων της ως τα μέσα του Μαρτίου για να παρακολουθήσει τη Μινούσκα την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινάει τώρα την ανάπτυξή της και άρα θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλη Μαρτίου. Αλλά ήδη έχουμε κληθεί να δώσουμε κάποιες ιδέες πιθανής, για την πιθανή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανάπτυξη για τις ε, σχετικές αποστολές των Εθνών και φαίνεται τα κράτη-μέλη να προτιμούν ή τουλάχιστον να αναλογίζονται το ενδεχόμενο μιας συμβουλευτικής αποστολής. Αυτή λοιπόν η ιδέα της διαχείρισης κρίσεων έχει ήδη ε, τύχη επεξεργασίας, έχει παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη και θα αναπατώ με αυτό συνέβη εχθές μόλις και εφόσον συμφωνήσουν να συνεχίσουν χωρίς εκτελεστική εντολή σε πιο μικρή ε, σύνθεση μπορεί να πάει στο Συμβούλιο το, της Αμήνης της 21 Δεκεμβρίου, αλλά δεν θέλω να προδικάσω τίποτα γιατί αύριο ξεκινάει το Συμβούλιο. Ε, για την έμπολα έγινε, για τον ιό έμπολα έγινε σύντομη συζήτηση. Καταγράφηκε κατάσταση σε ένα στιγμιότυπο, ούτως Έγινε επίσης εν συντομία συζήτηση για την πορεία εν ώψη των συστήσεων κυρίως του χρόνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας όπου είπατε εκπρόσωπος επιβεβαίωσε τη βούλησή της να αναλάβει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τα καθήκοντα που της έχουν αναδοθεί και να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο, μια στρατηγική αντίληψη, κάτι το οποίο ήδη έχει υποθεί βεβαίω, το επανέλαβε ωστόσο και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση με τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό και αν μπορεί να οδηγήσει σε μια επικαιροποίηση ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας ή όχι. Θα το δούμε αυτό. Είπατε εκπρόσωπος πάντως θέλει να τύχει προσεκτικής παρακολούθηση όλη η διαδικασία και να αναπτυχθούν συνεργικές δράσεις. Οι ε, δράσεις αυτές προβλέπεται να είναι όριμες τον Ιούνιο του 2015 για το Συμβούλιο. Πολλές φορές ζητήθηκε από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο να, από τους υπουργούς να υποβάλει μια έκθεση για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον Απρίλιο του 2015. για το επόμενο δηλαδή Συμβούλιο των Εξωτερικών, όπου όποτε φαίνεται θα είναι έτοιμη έκθεση. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις από τους υπουργού. Πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα πλαίσιο πολιτικής με πιο συστηματική αμυντική συνεργασία. Ένα από τα πολλαπλά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην υπατή εκπρόσωπο και τη σχετική υπηρεσία. Επίσης μια έκθεση για την κυβερνοάμυνα Έκτοτε έχουν επιβεβαιωθεί δύο ακόμα αποφάσεις οι οποίες είναι όριμες αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν από το Συμβούλιο, δεν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο ε, σε εκείνη τη συνεδρία επιφύλαξης κοινοβουλευτικής εξέλεξης Η εξέταση σημεία αφορούσε την Αταλάντη για το 2016. Επιβεβαιώνεται λοιπόν και μετά έχουμε μια απόφαση για την παράταση δραστηριοποίησης του Ευρωπαϊκού Λειτουργικού Κέντρου, Υπηρεσιακού Κέντρου, Επίσης ληφθεί απόφαση αυτή τη Δευτέρα. Η, παράταση, η, λειτουργία, η, επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης επίσης του επιχειρησιακού κέντρου, το οποίο πλέον θα καλύπτει και την περιοχή της Αχέλ και όχι μόνο το κέρας της Αφρικής. Η αναθεώρηση του μηχανισμού Αθηνά. Ε, πρέπει να έχει κρυθεί από το Συμβούλιο, αλλά δεν εξασφαλίστηκε αυτό, διότι δεν υπήρξε συνένεση. Συνεχίζουν τις συζητήσεις. Δύο-τρία θέματα μείνανε κρεμή. Συνεχίστε λοιπόν η δουλειά αυτή στο Συμβούλιο. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει άτυπα στη Ρήγα το Φεβρουάριο. Μια ευκαιρία ελπίζουμε για μια πιο στρατηγική συζήτηση των ε, προκλήσεων που συνεπάγονται οι βρυδικέ εχθροπραξίες που αφορά ιδιαίτερα και τον ΝΑΤΟ και το συζήτησαν και οι Υπουργοί των Εξωτερικών του ΝΑΤΟ εχθές. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σύντομη συζήτηση για τις μεθόδους εργασίας, γιατί είπα ότι εκπρόσωπος θέλησε να χαράξει ένα νέο δρόμο με άνοιγμα γιατί μίλησε προς τους Υπουργούς Αμήνης είπε ότι προσπαθεί να τους επισκέπτεται κάθε φορά που βρίσκεται σε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη το έχει πράξει με μια-δύο επισκέψεις θέλει δηλαδή να έχει καλύτερη χρήση των συναντήσεων με τους Υπουργούς Αμήνης δεν χρειάζεται να πολλαπλησιαστούν αυτές οι συνεδριάσεις αλλά να αξιοποιηθούν καλύτερα με καλύτερη διάρθρωση καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και η πρόθεση της υπάτησης εκπροσώπου είναι να αξιοποιήσει καλύτερα τις άτυπες δυνατότητες επαφής με πρώτη αυτή της Ρήγα και θα δει στη συνέχεια πώς θα έρθει σε επαφή με τους ε, υπουργούς στο πλαίσιο των επίσημων δομών της ε, κοινής Ασφάλειας και Σε Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ και περιμένω από τα μέλη τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους. Μπα, όχι, μάλλον είσαστε όλοι εξαντλημένοι. Ήταν και πολύ σαφής η παρουσίασή σας, κύριε Γενική Γραμματεύ. Σας ευχαριστούμε. Και περιμένουμε να σας ξαναδούμε την επόμενη φορά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να παραμένουμε ενήμεροι για τις εξελίξεις ε, του Υπουργείου των Εξωτερικών και στις δυο τους συνθέσεις. Ευχαριστώ θερμά. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, έτσι τελειώνουμε τις εργασίες μας για σήμερα. Προσεχή συνεδρίαση τον Ιούλιο, λέει ο Μιλήτρια, στις 21 του μηνός, μάλλον εννοεί τον Ιανουάριο. Και σας εύχομαι χρόνια πολλά. January, sorry. I'm tired. <laughs> I'm... ναι, με συγχωρείτε και εγώ κουρασμένη είμαι τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα να πούμε μόνο τον Ιούλιο. Λοιπόν, 21 Ιου... Ιανουαρίου και εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και θα τα ξαναπούμε τον Ιανουάριο.